Good morning. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Για να ξεκινήσουμε το δεύτερο τμήμα των εργασιών της Υποεπιτροπής ΣΕΝΤΕ. Πρώτο θέμα στη σημερινή μερίστη διάταξη είναι η ενημέρωση, οι υπηρεσίε πληροφοριών για την ανατολική γειτονική σχέση. Θα σας παρουσιάσουμε την περίπτωση της Μολδαβίας και με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τους εξαιρετικούς μας καλεσμένους, την κυρία Σουζάνε Κίφερ καταρχήν, πασίγνωστη σε εμά γιατί ήδη συμμετείχε σε συζητήσεις κατά το πρώτο ήμιση της κοινοβουλευτικής μας θητείας. Η κυρία Κίφερ εκπροσωπεί τη Stratcom East που ε, τη συνδράμει και η ΕΕΔ. θα εμπλουτίσει τις γνώσεις μας για στρατηγικές πληροφορίες και μάλιστα η Stratcom είναι τμήμα της ΕΕΔ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης Έχουμε μαζί μας και την κυρία Νατάλια Μωράρη, που είναι δημοσιογράφος από τη Μολδαβία και πρόεδρος της ε, πλατφόρμας ΜΜΕ με το όνομα Αλτερνατίβα ή Media Alternativa. Θα μας παρουσιάσει την κατάσταση στη Μολδαβία ε, σε ό,τι αφορά την κατάσταση αυτή στρατιωτική Επίσης είναι μαζί μας και ο κύριος Πέτρο Μακοβέη που είναι πρόεδρος ε, της ε, Μορδαβικής Ένωσης Ανεξάρτητο Τύπου. Αυτό το θέμα της ε, χρήσης των πληροφοριών ως εργαλείου πολεμικού είναι ένα θέμα που μας τράβηξε την προσοχή και μάλιστα έχουμε δράσει και πρωτοβουλίε τη ΥΠΑ τη εκπροσώπου Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε δράσεις και του Συμβουλίου μέσω των συμπερασμάτων του Συμβουλίου αλλά και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα αυτό είτε στην δική μας υποεπιτροπή είτε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων αλλά και σε άλλες επιτροπές. Χωρίς άλλη καθυστέρηση να δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Κίφερ, μετά στην κυρία Μωράρη και τέλος τον κύριο Μακοβέη. Κυρία Κίφερ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά θα σε ενημερώσω για, την, το πώς επηρεάζουν τα ξένα ΜΜΕ τη δημοκρατία της Μολδαβίας και τις δραστηριότητες ε, της ε, ομάδας κρούς, ομάδας εργασίας East Stratcom στη Βολδαβία. Καταρχήν, η ομάδα αυτή ιδρύθηκε το 2015 με στόχο να αντισταθμίσει και να διαψεύσει τις ε, επικοινωνιακές εξτρατείς της Ρωσίας στη Μολδαβία και μάλιστα είμαι ε, εκπρόσωπος της ΕΙΕΔ, γιατί η ίδια η ΕΙΕΔ σε αυτή την ομάδα εργασίας. Έχουμε μια ε, φευρία εντολή, αλλά πολύ ολιγομελή ομάδα. Καταρχήν κάποια στατιστικά στοιχεία που δείχνουν τον αντίκτυπο της δραστηριοποίησης των ε, ρωσικών ΜΜΕ στην δημοκρατία της Μολδαβίας και πώς επηρεάζουν την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Βέβαια, καταλήξαμε σε αυτά τα στοιχεία χάρη στη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, γιατί πολύ συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει δημοσκοπήσεις ε, στις χώρες Ανατολικής Γειτονίας και ως εκ τούτου έχουμε τη δυνατότητα να υπολογίσουμε το σχετισμό μεταξύ της κατανάλωσης των μέσων των ρωσικών ΜΜΕ και των εντυπώσεων της εικόνας που έχει στις χώρες Ανατολικής Γειτονίας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χρήστες ε, των ε, ρωσικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στη Μολδαβία έχουν λιγότερο καλή ε, εντύπωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μάλλον αρνητική γνώμη τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα οι χρήστε των ε, ντόπιων μέσων μαζικής ενημέρωσης αντίθετα έχουν πολύ θετική γνώμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα έχουν ακόμη και καλύτερη γνώμη από ό,τι στις χώρες μέλη. και είναι λίγοι αυτοί που έχουν αρνητική γνώμη. Σε καμία άλλη χώρα της Ανατολικής Γειτονίας δεν ε, είδαμε την σημαντική επιρροή που έχει η χρήση, η παρακολούθηση των ρωσικών ΜΜΕ για το κύρος και την υπόλοιψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε μια χώρα. Στις άλλες χώρες της Ανατολικής Γειτονίας, στην Γεωργία για παράδειγμα ή την Ουκρανία, εκεί ε, έχουμε χαμηλότερη παρακολούθηση των ρωσικών ΜΜΕ, ενώ στη δημοσκόπηση αυτή 61% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι παρακολουθούν ρωσικά ΜΜΕ. Οπότε διαπιστώνουμε ότι η διείσδυση των ρωσικών ΜΜΕ στη Μολδαβία είναι υψηλή και επηρεάζουν αρνητικά το κύριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη χώρα. Με αποτελέσματα αυτά τα αρνητικά στη δημοσκόπηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω καταρχήν ποια στρατηγική οθετήσαμε για να αντικρούσουμε αυτή την πολιτική. Συνεργαζόμαστε από τον Ιανουάριο του 2016 με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και η στρατηγική μας είναι ως πρώτο βήμα καταρχήν να αυξήσουμε και να κάνουμε πιο αποτελεσματική την επικοινωνία μας ε, ε, για το πώς βοηθούμε τη Μολδαβία ως Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθούμε να βρούμε πιο αποτελεσματικά μέτρα σε πλήρη συνεργασία με την αντιπροσωπεία μας και τη Γενική Διεύθυνση ΝΙΕΡ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να φτάσει το μήνυμα στο ακροατήριο. Έχουμε ενισχύσει τη διαδικτυακή μας παρουσία και ε, έχουμε πιο στοχευμένες δράσεις στη χώρα αυτή. Βέβαια δεν ήταν προτεραιότητα μας η παραπληροφόρηση που γίνεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μολδαβία. Γιατί μετά τις τελευταίες έρευνες ε, για τη διάψευση των fake news ε, διαπιστώσαμε ότι αν έχουμε ένα ακροατήριο που πιστεύει σε αυτό το μύθο, σε αυτή την ψεύτικη δήλωση, τις ανακριβείς ειδήσει, ε, έδειξαν οι έρευνες ότι είναι πιο αποτελεσματικό το να επικεντρωνόμαστε στα δικά μας μηνύματα, από το να αναλωνόμαστε, στο να διαψεύδουμε τις ανακριβείς ειδήσει που κυκλοφορούν. Πιο αποτελεσματικό είναι να προσπαθούμε να μεταδώσουμε το δικό μας μήνυμα. Να σας παρουσιάσω τις τρεις εκστρατείες ε, που είτε είχαμε είτε ε, δρομολογούμε στη Μολδαβία, προσπαθώντας να περάσουμε το δικό μας μήνυμα, να επικοινωνήσουμε σωστά το δικό μας μήνυμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη εκστρατεία είναι να συμπαρασταθούμε και πάλι και να εμπλακούμε στην ε, καταπολέμηση της διαφθοράς, γιατί στη Μολδαβία οι πολίτες πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε ε, διεφθαρμένους πολιτικούς ή όχι αδιάφθορους, σε πάση περιπτώσει, και μάλιστα ε, η οχι αδιαφθορους σε παση περιπτωσει και μαλιστα η εξτρατεια μας συνέπεσε και με το πρωτάθλημα το ποδοσφαιρικό. Εκεί είχαμε την εκστρατεία κόκκινη κάρτα στη διαφθορά. Προσκαλέσαμε και κόσμο και μάλιστα στην Κισινάου ε, ε, είχαμε μία συνέντευξη με έναν διετή που είπε ακόμη και όταν φίλοι του παίζουν ε, δεν το λαμβάνει υπόψη. Και προσπαθήσαμε αυτό το μήνυμα να το περάσουμε και στα ποδοσφαιρικά γήπεδα και γενικώ στον κόσμο. Συνεργαζόμαστε επίσης και με ΜΚΟ που ενεργοποιούνται στην πάταξη διαφθοράς και μας ε, μιμήθηκαν και πολιτικοί, κάτι που δείχνει πόσο σωστή ήταν η προσέγγιση μας και εύστοχη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, ε, δεύτερη εκστρατεία μας, που διεξήχθη μεταξύ Οκτωβρίου του 2016 και Ιανουαρίου του 2017, εκεί από κοινού με την αντιπροσωπεία βρήκαμε ανθρώπους που η ζωή τους είχε αλλάξει χάρη στην Ευρωπαϊκή Συνδρομή στην Μολδαβία και σε σύντομα βιντεάκια Ε, παρουσιάσαμε το έργο τους ε, μέσω αυτής της κοινωνικής διαφήμισης ε, και πέντε ή έξι τηλεοπτικά κανάλια μετέδωσαν αυτά τα βιντεάκια και μάλιστα το, η ακροματικότητά τους και το μερίδιο τους στην αγορά ΜΜΕ ήταν δύο τρίτα της συνολικής αγοράς. Επίσης, σε μια έρευνα που κάναμε ποσοτική διαπιστώνουμε ότι αυτά τα βιντεάκια πραγματικά είχαν απήχηση γιατί προβάλλονταν πολλές φορές τη μέρα σε πολλά τηλεοπτικά κανάλια, κάτι που έφτασε στον κόσμο. Επίσης, ε, ετοιμάζουμε τώρα μια εκστρατεία για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όσοι παρακολουθούν το πολιτικό σκηνικό στη Μολδαβία γνωρίζουν ότι υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και κυρίως για τη σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου ήδη έχουμε ξεκινήσει ε, την εκστρατεία μας για να ενημερώσουμε τον κόσμο για το μέγεθος των εμπορικών συναλλαγών γιατί ο κόσμος έχει εσφαλμένη εντύπωση για το μέγεθος αυτών των συναλλαγών και επίσης δείχνουμε ε, επιτυχημένε εταιρείε που εξάγουν προς την ευρωπαϊκή αγορά και ε, θα ξεκινήσουν από την επόμενη Κυριακή τις, ε, τις σχετικές πρωτοβουλίες. Επίσης έχουμε quiz, συνεντεύξεις τύπου, συνεντεύξεις με επιτυχημένους επιχειρηματίες. Βλέπετε εδώ τις δραστηριότητες προβλέπουμε ώστε να προβάλλουμε τα πλεονεκτήματα της συμφωνίας αυτής ελεύθερων συναλλαγών και να την προβάλλουμε ως βάση για την ευημερία της ε, μολδαβικής κοινωνίας. Αυτά σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι έτοιμη να απαντήσω σε απορίες. Ευχαριστώ την κυρία Κίφερη. Η κυρία Μωράρη έχει το λόγο. Καλημέρα σε όλους. Ε, ζητώ συγγνώμη εκ προημίου γιατί τα αγγλικά μου δεν είναι τόσο καλά. το να πούμε ότι δεν είναι πολύ θετική η κατάσταση στη Μολδαβία ε, είναι σχεδόν το να κάνουμε λάθος. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην κατάσταση της αγοράς. Όταν έχουμε ένα απόλυτο μονοπόλιο με πολιτικό συμφέρον, η ανάμειξη αυτή καθιστά τα πάντα απολύτως δυνατά. Έχουμε λοιπόν μονοπωλιακή μεταχείριση των μέσων ενημέρωσης, η οποία σχετίζεται με το πρώτο αίτιο της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα. Εγώ είμαι ρωσόφωνη Μολδαβή, αλλά όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την ρωσική κουλτούρα, το ρωσικό πολιτισμό και τη γλώσσα στη χώρα μας που είναι σημαντικά, αλλά με μια εκστρατεία παραπληροφόρησης και ξεκινώ με κάποια μεγέθη. Στην αγορά του τύπου μέχρι το 70% όλου του περιεχομένου του τηλεοπτικού προέρχεται από την ρωσική τηλεοπτική αγορά. δεν είναι υψηλά ποιοτικό, αλλά είναι φθηνότερο και είναι πάρα πολύ ε, σύνηθες για το κοινό στη Μολδαβία, γιατί είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό. Και όλοι οι σταθμοί είτε είναι άμεσα είτε έμεσα συνδεδεμένοι με τους μεγάλους ομίλους, ο μεγαλύτερος από τον Βλάντμπαχ Χονιούκ και ο δεύτερος ε, που είναι συνδεδεμένος με τον Ίγκορ Ντόντον. Δεν είναι άμεσα ιδιοκτήτης του ομίλου αυτού, αλλά είναι μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος ο πρόεδρος του και φίλος του επίσης μέλος του Κοινοβουλίου. Έχουμε λοιπόν την Nova TV, το κανάλι αυτό, και τα δύο μεγαλύτερα κανάλια ελέγχουν το 85% όλης της διαφημιστικής αγοράς. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της ενώσεως ανεξάρτητου τύπου, ο συνάδελφος είναι εδώ και θα σας το πει, η Μολδαβία έχει πλημμυριστεί από ρωσικά blog και show καθημερινά μέσω των δύο αυτών τηλεοπτικών σταθμών. Μέσα τα οποία ενημερώνουν τον τρόπο τον οποίο η Ρωσία διαδραματίζει θετικό ρόλο σε όλα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή και γιατί η Ρωσία είναι θύμα των ΗΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα κακά στην περιοχή συμβαίνουν λόγω ημών με ύψιλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ κτλ. Μας πληροφορούν, μας πληροφορούν επίσης σχετικά με την ηθική κατάπτωση της δύση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής και ο κύριος Πούτιν είναι ο μόνος υπερασπιστή της ελευθερίας. Ο ρωσικός σταθμός πέρα κανάλ, αν ακούσαμε καλά, με ιδιαίτερα επιθετική εκστρατεία τύπου. Ο ιδιοκτήτης του είναι ο Βλάτπαχ Κονιούκ, με συγχωρείτε, ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος μας ε, ενημερώνει καθημερινά για τις ερωαϊκές του αξίες, αλλά ταυτόχρονα μας ενημερώνει μέσω των blog και των talk shows στα κανάλια του για την κατάπτωση, την ηθική κατάπτωση της δύσεως. Εδώ θα σταματήσω με την τηλεοπτική προπαγάνδα και θα περάσω σε εκείνη του διαδικτύου που είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικό πρόβλημα. Και να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Δύο όμιλοι, οι διοικητές των οποίων είναι η Ικονίου και τον Τόν και πάλι, ε, έχουν προχωρήσει σε μια εκστρατεία παραπληροφόρηση σχετικά με τους μετανάστες από τη Συρία και εκφράζουν ανησυχίε σχετικά με την εισβολή των Σύριων στην Μολδαβία σε περίπτωση που συγκεκριμένος υποψήφιος γινόταν πρόεδρος. Τα περισσότερα από τα μέσα αυτά αν επανεκπέμπουν στην ουσία ρωσικό περιεχόμενο. Επίσης έχουμε μία επιρροή στις εκλογές αν δείτε όλες τις εκθέσεις που έχουν υποβληθεί από ανεξάρτητους, ε, ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, βλέπουμε όλα αυτά αποτυπώνουν το ίδιο ε, επίπεδο ε, επιρροής και διαφοράς. Ελαμβάνουν εντολές από τους συναδέλφους τους στη Ρωσία, λέει ο Μιλήτρια, για το πώς θα διεξαγάγουν την προπαγάνδα αυτή και πολύ συχνά είναι ταυτόσιμη η προπαγάνδα που γίνεται στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο. Επομένως καθημερινά βομβαρδίζεται η Μολδαβία με παραπληροφόρηση από την ρωσική προπαγάνδα. Πώς θα μπορούσε ο, ο ελεύθερος τύπος να επιβιώσει υπό τις συνθήκες αυτές. Είναι σχεδόν αδύνατον όταν έχουμε μόνο το 15% του μεριδίου στην αγορά διαφημίσεων και υπάρχουν αρκετοί σταθμοί και μέσα ελεύθερου τύπου, λέει η ομιλήτρια. Το τοπικό περιεχόμενο ε, υποστηρίζεται ε, έντονα από το σύστημα του μονοπωλίου. Εάν κανείς ανήκει στους δύο μεγάλους ομίλους είναι παίκτη, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν επικρίνει την κυβέρνηση ή ότι έχει άμεση οικονομική στήριξη από τη Ρωσία. Το πολιτικό καρτέλ που οικοδομείται αυτή τη στιγμή μεταξύ των κυρίων Ποχοτνιού και ε, είναι παρόν στην αγορά και έχουμε το παιχνίδι του καλού και του κακού αστυνομικού που διαδραματίζουν αυτοί οι δύο και οι σταθμοί τους ε, ένα λάξ. Όμως έχω κάποια δυσάρεστα νέα. Μερικές φορές η ελεύθερη αγορά αρέσκεται στη διαχείριση μονοπωλίων και η Μολδαβία είναι ένα καλό παράδειγμα. Έχουμε τον άμεσο έλεγχο του 65% μέσω των ομιλών αυτών τη διαφημιστική αγορά, από κρατικού μάλιστα φορεί, και μπορεί κανείς να προχωρήσει μέχρι και 80% έκπτωση για καλούς πελάτες υπό την προϋπόθεση ότι όλο το περιεχόμενο θα διοικητευθεί μέσω των συγκεκριμένων αυτών ομίλων. Αυτό είναι ο τρόπος τον οποίο λειτουργούν και αυτό είναι ο, ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλίσει κανείς ότι δεν θα υπάρχει ελευθερία του τύπου για τους σταθμού που προσπαθούν να επιβιώσουν. Και δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι οι επιχειρήσει δεν θα ήθελαν να έχουν το 80%. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το, τα υψηλά ποσοστά ακροαματικότητος, το καλό business δηλαδή, και οι πόροι, η στήριξη που θα λάβουν. Δίνουμε μάχη για ένα εκατομμύριο ευρώ αξίας αγορά διαφημιστική όλη η σταθμοί που είναι ελεύθερη, το οποίο είναι ένα αστείο ποσό. Θα μπορούσε να μιλάει κανείς για πάρα πολύ καιρό για την αλλαγή της νομοθεσίας, αλλά στην ουσία αν υπάρχει βούληση μπορεί κανείς να αναλάβει δράση αμέσως. Πριν από δύο χρόνια το TV7, σταθμός που δουλεύω εγώ, έλαβε μια σημαντική απόφαση κατά τη διάρκεια του, του, Ουκρανικού πολέμου. Αποφασίσαμε να αλλάξουμε όλα τα ρωσικά blog και να αντικαταστήσουμε με τοπικά, με δικά μας πολιτικά show αναλύσεων μετά από αυτό χάσαμε σε ακροματικότητα, χάσαμε σε μερίδιο διαφημίσεων και μέχρι το τέλος του 2015 διεκόπη η άδεια μεταδόσεων που είχαμε και παραχωρήθηκε σε άλλο σταθμό συνεδεμένο με τον ε, Ίγκορ Ντοντών. Ενώ οι σταθμοί του κυρίου Ποχοτνούκ δίνουν άδεια στον MTVA της Μολδαβίας και αυτό που προκύπτει από αυτό είναι ότι η, ρωσικά, η ρωσική προπαγάνδα δεν είναι απλώς ένα πολιτικό μέσο εργαλείο, αλλά είναι ένα σύστημα οικονομικής εκμετάλλευσης. Αυτό που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να υποστηρίξει άμεσα τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Το οποίο συμβαίνει ήδη για Καλή ποιότητα μέσα ενημέρωση συμπεριλαμβανομένου του δικού μα στη Μολδαβία, του TV7. Και πρέπει να αναφέρουμε ότι το 80% των Μολδαβών χρησιμοποιούν τηλεόραση ως πρώτο μέσο ενημέρωσης. Αλλά έχουμε ένα διαφορετικό κόστος από τον, τα έντυπα ή άλλα, ε, άλλα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων στη Μολδαβία που καθημερινά ανοίγουν την τηλεόρασή τους και μέσω αυτής παρακολουθούν διάφορα, ε, διάφορες πολιτικές εκπομπές και τόξο. Ε, ε, εάν θέλουμε λοιπόν να ενημερώνεται αντικειμενικά το κοινό στη Μολδαβία, Πρέπει όχι μόνο να παρακολουθεί τι γίνεται με την αγορά των μέσων ενημέρωση, πρέπει να αναλάβει κανεί δράση άμεσα αυτή τη στιγμή. Thank Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάκοβεϊ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή να εκφράσω την απόψή μου σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην ε, Μολδαβία και στο μολδαβικό τύπο και ειδικά σε ό,τι αφορά την προπαγάνδα και την, το εργαλείο της προπαγάνδας. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω στα ρουμανικά. We have translation, yes? Yeah. Doamnelor și domnilor, atunci când vorbim despre Republica Moldova, trebuie să κατάσταση σε ό,τι αφορά τη Μολδαβία εμπεριέχει πάρα πολλού παράγοντε, γεωγραφικού παράγοντε, ιστορικού παράγοντε αλλά και γλωσσολογικού παράγοντε. Όλα αυτά λοιπόν στην σύνθεση του καταδεικνύουν ότι βρισκόμαστε ακόμα στην σφαίρα επιρροή τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η Μολδαβία λοιπόν είναι πρώην Σοβιετική Δημοκρατία και επί 70 χρόνια υπήρχε μια διαδικασία αποκρατικοποίησης, μια απόπειρα να αποδεχτεί στον κόσμο την είναι σλαβικής προέλευσης, αλλά ουσιαστικά ο κόσμος είναι ρουμανικής προέλευσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο επί όλης της ε, κυριαρχίες της Σοβιετικής Ένωσης ε, προσπάθησαν να πείσουν ε, τους Μολδαβούς Προσπαθούσαν λοιπόν να του πείσουν ότι είναι κυριλική ε, προέλευση ε, η μολδαβική γλώσσα. Είναι και τεχνητή γλώσσα και η ρουμανική γλώσσα είναι η ίδια γλώσσα, τα ρουμανικά με τα μολδαβικά. Αυτό ήταν αυτό που προωθούσαν. Φυσικά είναι σφάλμα αυτό και λάθο. Ε, επί σειρά λοιπόν ετών προσπάθησαν να πείσουν την μολδαβική, το μολδαβικό λαό για τα πράγματα αυτά. Αυτά δεν μπήκαν και στο Σύνταγμα σε κάποια στιγμή. Και αυτό πραγματικά είναι κρίμα, γιατί είναι κάτι το οποίο το, το χρησιμοποιεί τώρα και ο πρόεδρο τη Μολδαβική Δημοκρατία. Το πρώτο λοιπόν που κάνει, έκανε όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του είναι ότι άλλαξε το επίσημο όνομα της γλώσσας μας από ρουμάνικα σε μολδαβικά. Το 1991 λοιπόν η υπερτινιστερία στην Ευρωτερία ξέσπασε πόλεμο και η Ρωσική Ομοσπονδία άμεσα παρενέβη και μετά από 26 χρόνια Πλέον αυτό το θέμα δεν το ελέγχουν ακόμα οι μολδαβικέ αρχέ. Είναι λοιπόν εξαιρετικά ασταθή η κατάσταση και αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Μία περιοχή στο νότο Μια περιοχή λοιπόν στην Νότο η οποία είναι υπέρ τη ρωσική επιρροή. Η ρωσική επιρροή πρέπει να ξέρετε είναι πάρα πολύ έντονη στη Μολδαβία και αυτό διατυπώνεται με, διάφορους, με διάφορες μεθόδους. Υπάρχουν διάφορες πηγές προπαγάνδας σήμερα από τη Ρωσία, οι οποίες άσκουν επιρροή και στον πρόεδρο. Έχουμε την νομοθεσία του πρόεδρου στο και σε ό,τι αφορά την ε, προσπάθεια να διακοπεί η συνεργασία της Μολδαβίας με τον ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά λοιπόν γιατί υπήρξαν αιτιάσει σε ό,τι αφορά μάλλον την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ κυρίως από ρωσικές πηγές. Και όλα αυτά λοιπόν είναι απίστευτα. Απίστευτα για κάποιον και για ένα έθνος το οποίο μπορεί πραγματικά να ζητήσει πραγματικές πληροφορίες. Θα πρέπει λοιπόν ο ίδιος ο κόσμος να ασκήσει πίεση, γιατί πολλοί κόσμος έχει εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης και στη Ρωσική Ομοσπονδία. Τα τοπικά μέσα, το είπε και ο συνάδελφος, είναι υπό την ε, ε, πίεση και υπό την επιρροή των πολιτικών. Ακριβώς λοιπόν το ίδιο έκαναν διέδωσαν αναλυτικές πληροφορίες, μετά έγιναν και οι και το Συμβούλιο των Μέσων που είναι η ρυθμιστική αρχή στον τομέα αυτό ε, επέβαλε ποινές. Ε, οι εκπομπές ε, όμως αυτές δεν διαψεύθηκαν. Δεν βγήκαν οι σταθμοί να διαψεύσουν τις πληροφορίες που διαδόσαν. και φυσικά η ρωσική επιρροή ασκείται και από τους πολλαπλούς ρωσικούς σταθμούς που μεταδίδονται στη Μολδαβία από, τοπικές, από τοπικούς φορούς και πρόκειται για μεταβιβάσεις οι οποίες δεν ε, ελέγχονται από τους τοπικούς ε, και τους εθνικούς νόμους. Δεν τα ελέγχει δηλαδή όλα αυτά το Σχετικό Συμβούλιο Οπτικοδοτικών Μέσων και την προπαγάνδα που ασκείται. Θα ήθελα να την περιγράψω, αλλά να σας υπενθυμίσω πρώτα ότι η ρωσική περιοχή αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα και ύστερα υπάρχει και η Ορθοδόξη Εκκλησία, πάρα πολύ σημαντικό φορέας και αυτός. Έχουμε δύο Μητροπόλεις, η Μολδαβική ε, Μητρόπολη και η Μητρόπολη της Βεσαραβίας υπό το Ρουμανικό Πατριαρχείο. Εκεί λοιπόν πραγματικά Υπάρχουν ε, πράκτορες οι οποίοι είναι υπέρ της Ρωσίας. Τα τελευταία δέκα χρόνια στη χώρα μας υπήρξαν εξελίξεις και σε όλες τις ε, εκλογικές αναμετρήσεις, ο κλήρος και η Μολδαβική Μητρόπολη πάντα υποστηρίζει τους Ρώσους υποψηφίους, ανεξάρτητα από το κατά πόσον ήταν υποψήφιοι από το Κομμουνιστικό ή το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ο πρόεδρος τη της Δημοκρατίας βασίζεται και προασπίζει τις χριστιανικές αξίες ε, στη χώρα μας. Το 2006 στις προεδρικές εκλογές ε, οι εκπρόσωποι του κλήρου διέδωσαν αναλυθείς ε, πληροφορίες οι οποίες ήταν και αιτιάσεις και κατηγορίες κατά κάποιων υποψηφίων. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε αντίπινο, οποιαδήποτε συνέπεια. Το Κοινοβούλιο τελικά έλαβε ένα έγγραφο για την αλλαγή του σχετικού νόμου προκειμένου να μην μπορούν να ασκούν οι εκπρόσωποι του κλήρου της Εκκλησίας τέτοια προεκλογική προπαγάνδα. Αλλά αυτό δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί στην πράξη, παρόλο που υπάρχει σχετική υποχρέωση για εφαρμογή του νόμου αυτού μέσα σε τρει μήνες, Ένα άλλο παράγοντα επιρροή είναι προφανώ και τα κοινωνικά δίκτυα, προσφάτως, αλλά και τα website, οι ιστοσελίδες. Υπάρχει ο κόμβος Sputnik, ε, που στην ε, Δημοκρατία της Μολδαβίας αποτελεί πλέον ε, μια υπηρεσία τύπου. Και πρέπει να πούμε όμως ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κατάρτισης των δικών του συντήσεων. Και το σχετικό Συμβούλιο Οπτικοακουστικών Μέσων πολύ διαπιστώνουμε δυστυχώ ότι δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά του και δεν επιβάλλει και τι σχετικέ κυρώσει που προβλέπουν. Την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, η δική μου ένωση υπέβαλε μία έκθεση παρακολούθηση για πέντε ρωσικού σταθμού, οι οποίοι εκπέμπουν μέσω τοπικών σταθμών LTRN, RANDEVER, STS και NTV μεταξύ άλλων. Όλοι λοιπόν σχετικά αυτοί οι σταθμοί, όλοι σχεδόν αυτοί οι σταθμοί, αποτυπώνουν την εντατικότατη προπαγάνδα από πλευρά της Ρωσίας. Και αυτά λοιπόν εκπέμπονται στο εσωτερικό της Μολδαβία. Πάντα με το ίδιο θέμα. Ό,τι κακό συμβαίνει και στραβώσει τον κόσμο, το έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΠΑ ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Η Ρωσία, από την άλλη, είναι ο πυλώνας ε, της, ε, του πολιτισμού και προσπαθεί να σώσει τον κόσμο από την Αμερικανική επιρροή. Αυτό είναι το μήνυμα που μεταδίδεται. Δυστυχώ, η Ρωσία δεν εκτιμάται αρκετά στην παγκόσμια κοινότητα μετά από όλα αυτά που έχει συνδράμει. Γιατί είναι εξαιρετικό ο ρόλο της Ρωσική Ομοσπονδία και εξαιρετικό ο ρόλος του Πούτιν ως ε, πολέμιος της τρομοκρατίας και πιστός προασπιστής ε, της δημοκρατίας και του χριστιανισμού. Αυτά είναι τα μηνύματα τα οποία προβάλλονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δε ε, υπονομεύει τις αξίες αυτές και αποτελεί αρνητικό παράγοντα και το ΝΑΤΟ ουσιαστικά αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και στην στρατιωτική παρέμβαση. Το μεγαλύτερο δε τμήμα των μηνυμάτων που περνάνε μέσα από την προπαγάνδα της ρωσικής τηλεόρασης απευθύνεται προφανώς στα θέματα της Ουκρανίας. Η ρωσικοί λοιπόν σταθμή δεν ασχολούνται σχεδόν καθόλου με τα εσωτερικά του ζητήματα. Εξετάζεται λοιπόν η κατάσταση στην ε, Ουκρανία, στα διάφορα μέσα ενημέρωση, σε διάφορα talk show, εκπομπέ. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο αυτό και υπάρχει για παράδειγμα το εξή μήνυμα ότι η Ουκρανία όπου να είναι θα διαλυθεί. Ένα άλλο μήνυμα το οποίο προβάλλεται είναι ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζεται στην Ευρώπη ως ε, χώρα δεύτερης κατηγορίας και κάτι άλλο να σας αναφέρω. Είδαμε στο RNTV ε, κάποιες συγκεκριμένες εικόνες. Εικόνες που αποτυπώνουν νέους ανθρώπους δίπλα στο Mannequin Peace στις Βρυξέλλες. Με ένα ποτήρι νερό και ο συντονιστή τη εκπομπή ε, ε, βγήκε και είπε ότι κοιτάξτε έτσι αντιμετωπίζουν και του Ουκρανούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, σαν να του ποτίζουμε δηλαδή ε, ούρα τους Ουκρανούς. Αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο προσπαθούσαν να περάσουν. Το υποτιμητικό αυτό μήνυμα, ότι οι Ευρωπαίοι δηλαδή τάχα θέλουν να ε, να αλλάξουν ακόμα και την οτροπία των παιδιών των ίδιων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ουκρανία. Τους διδάσκουν δηλαδή παιχνίδια σατανικά. όπου ανοίγουν ε, τα σωθικά των ανθρώπων και τους δείχνουν τέτοια μηνύματα. Ε, μηνύματα τα οποία, ξέρετε, κάνουν ε, συγκρίσεις ε, Ό,τι κακό και στραβό λοιπόν στον κόσμο είναι από τη ΣΥΠΑ. Και ό,τι καλό και ευγενέ από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτά τα μηνύματα, ξέρετε όμως, συστηματικά μεταδίδονται. Πρόκειται για προπαγάνδα καθημερινή και πολύ συστηματική. Και υπάρχουν πάρα πολλέ ε, τεχνικές και μέθοδοι για την προπαγάνδα αυτή. Μονομερής παρουσίαση όλων των γεγονότων, κλιμάκωση τη προπαγάνδας, ε, ε, υπόγεια, ύπουλα, μηνύματα και πολλοί άλλοι, πολλές άλλες μέθοδοι. Και έγιναν και πάρα πολλές συζητήσεις σχετικά. Διάφορα μηνύματα και αιτιάσεις, ε, δρυμία, κατηγορώ τα οποία δεν έχουν να κάνουν όμως απαραίτητα με το θέμα το οποίο συζητιέται και πρόκειται για έτσι ύπουλα ε, μηνύματα, τα οποία ε, υπόγεια μεταβιβάζονται, κάτι άλλο, για την Ουκρανία και τους τρομοκράτες, για παράδειγμα. Ουκρανοποίηση. Ε, τέτοια μηνύματα τα οποία μεταβιβάζονται στους ακροατές. Ύστερα διάφορες καρικατούρες, διάφορες, ε, διάφορα κόμικ, διάφορα κινούμενα σχέδια τα οποία διακομωδούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς εξυμνούν την Ρωσική Ομοσπονδία. Επίσης, στην Δημοκρατία της Μολδαβίας υπάρχουν και ενημερωτικοί κόμποι, κάποιοι από τους οποίους χρηματοδοτούνται από τη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά και από επιχειρήσει αντιστοιχώ. Ε, ε, προφανώς λοιπόν προβάλλουν το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση να, να όπου να διαλύεται. Ότι ε, έχει κηρυχθεί πόλεμος ε, με την Ρωσία και το ίδιο κάνει και η Μολδαβία και άρα η Μολδαβία θα έχει την ίδια τύχη με την Ουκρανία αν δεν ακολουθήσουν οι Μολδαβοί πολιτικοί την οδό της Ρωσίας ε, προφανώς και ότι αυτό θα ήταν προφανώ καταστροφικό για τη Μολδαβία και το καθεξή. Μόνο ειδήσει λοιπόν. Δηλαδή η Δύση ευθύνεται για όλα τα προβλήματα της Μολδαβίας και το μόνο που μπορεί, ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει είναι η Ρωσία. Προβάλλεται επίση το μήνυμα ότι δεν θα ε, εορτάζεται πλέον η επέτειο τη 9η Μαου στη Μολδαβία ω επέτειο ανεξαρτησία. Γιατί πάντα υπάρχει μία αντιπαλότητα Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κατά τη Ρωσία. Ε. Και πάντα γίνεται απόπειρα υπονόμευση τη Δύση. Προβάλλεται επίση το μήνυμα ότι όσοι πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ενωποίηση είναι αφελεί μέχρι και ηλίθιοι. Και διαρκώ κατηγορούνται και ενοχοποιούνται όλοι οι, άνθρωποι ε, κατά διαστολή. Υπάρχουν οι καλοί, υπάρχουν οι κακοί, υπάρχουν οι αθώοι, υπάρχουν και οι ένοχοι. Και προφανώς αυτό προβάλλεται και στα talk shows, στις συζητήσεις, καλούνται ε, εμπειρογνώμονες οι οποίοι υποστηρίζουν θέσεις υπέρ του Κρεμλίνου και μάλιστα με πολύ μαχητικό τρόπο. Βρίζουν, οι άλλοι δε, οι οποίοι διακηρύττουν κάτι αντίθετο, δεν τους αφήνουν καν να μιλήσουν. Και οι συντονιστέ ε, των εκπομπών και αυτοί επιλέγονται επί τούτου, προκειμένου να προωθούν ακριβώς τα συμφέροντα αυτά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρή η κατάσταση η οποία χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή τη δημοκρατία της Μολδαβίας. Υπάρχει και ε, ένα website, μια σελίδα μια εφημερίδα της ε, Μολδαβίας, όπου δημοσιεύτηκε προσφάτως ένα άρθρο, το οποίο αναφέρει ότι όσοι μιλούν ρωσικά στη χώρα να κάτσουν να πεθάνουν και να μην ε, τους δίνουμε ούτε καν φάρμακα στα φαρμακιά. Μα όλα αυτά είναι ψέματα. Δεν υπάρχει τέτοια διακρατική μεταχείριση στην ε, δημοκρατία της Μολδαβίας. Όλα αυτά στο σύνολο τους ε, συνθέτουν ένα μεγάλο κύμα παραπληροφόρησης, παραπλάνησης, προπαγάνδας στο γραπτό, τον εντυπωτύπο, στα κοινωνικά δίκτυα, στην τηλεόραση, στο ράδιο. Όλα αυτά λοιπόν ως κύμα πληροφοριών είναι απεχθή. Και δυστυχώ στη Δημοκρατία τη Μολδαβία στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάποια συντονισμένη στρατηγική για την προστασία της πληροφόρηση. Μία στρατηγική, για παράδειγμα, για την ασφάλεια του τύπου. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία θα μπορούσαν να αφορούν την προστασία της ε, πληροφόρησης προκειμένου να είναι σωστή και δίκαιη. Και εγώ και οι συνάδελφοι έχουν παρουσιάσει αυτή την κατάσταση και κάποιοι πολιτικοί δε στην δημοκρατία της ε, Μολδαβίας έχουν και αυτοί συμφέροντα να προβάλλονται τα ρωσικά μηνύματα, οι ρωσικοί σταθμοί και πώς ε, να αντισταθούν σε αυτούς. Θεωρούμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ασκήσει πίεση στις Μολδαβικές Αρχές και να δώσει και ενδεχομένω και αρρωγή και χρηματοοικονομική, χρηματική βοήθεια για να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία θα είναι και μετρήσιμα. Και στον τομέα της ενημέρωσης η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει με διάφορους τρόπους την δημοκρατία της Μολδαβία, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την διεξαγωγή μεταρρυθμίσεων και γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μολδαβική κυβέρνηση για να υπάρξει συγκεκριμένη πρόοδος και στα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να αναπνεύσουμε λίγο από την προπαγάνδα αυτή και, από την εξωτερική προπαγάνδα, αλλά και κυρίως από την εσωτερική προπαγάνδα, την οποία ανέφερε και η συνάδελφος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να απαντήσω στις ερωτήσεις σας εφόσον υπάρχουν. Thank you. Σας ευχαριστούμε. Περάμε στη συζήτηση. Ο κύριος Γκάλερ ζήτησε το λόγο πρώτα. θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί έφτασα καθυστερημένα στη συνεδρίαση και δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω από την αρχή όλες τις ομιλίες. Ελπίζω να υπάρχει και κάποιο έγγραφο, κάποιο υλικό γραπτό για να ενημερωθούμε. Ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή είμαστε απασχολημένοι με την δημοσιονομική διαδικασία ε, και προσπαθούμε με τον προπολογισμό να στηρίξουμε και τη στρατηγική μας ε, επικοινωνιακή πολιτική. Και διαπιστώνω ότι η κατάσταση είναι διαφορετική στα κράτη-μέλη. Εκεί υπάρχουν μονάδες ή οργανισμοί, διάφοροι φορείς που προσπαθούν να αντικρούσουν αυτή την ε, πολιτική παραπληροφόρηση. Είναι δυνατή η διασύνδεση, η ανταλλαγή πληροφοριών για να μην είναι ο καθένα στη γωνιά του απομονωμένο ε, ε, και να υπάρχει διασύνδεση. Βέβαια, από το Κρεμλίνο εκπορεύεται μία ενιαία στρατηγική ε, ενάντια όλων μας. Αλλά εμείς μπορούμε να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητά μας με καλύτερη συνεργασία, με διασύνδεση μεταξύ των φορέων που ασχολούνται με αυτό το θέμα της καταπολέμησης παραπληροφόρησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Φροντζούλικα. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τους τρεις καλεσμένους μας για την παρουσία τους και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Μακοβέη που μας παρουσίασε την πραγματικότητα για το τι πραγματικά συνέβη στη δημοκρατία της Μολδαβίας. Στη χώρα αυτή και ο λαός της Μολδαβίας, όπως όλοι ξέρετε, από την ιστορία του, την ε, παράδοση, την τις παραδόσεις τους, την ιστορία τους. Ε, ε, είναι τμήμα της Ευρώπης, είναι τμήμα της νοτιοανατολικής Ευρώπης η Μολδαβία και ο λαός της Μολδαβίας. Θα πρέπει σε αυτή την... αυτό το πλαίσιο να επιστρέψει η Μολδαβία. Και όταν εξετάζουμε την κατάσταση Μολδαβία, να δούμε πού ανήκει, στη Δύση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ανατολή με, την, ε, ε, με τη Ρωσία ή με τις ε, ευρασιακές οργανώσεις. Είναι θέμα και πολιτικής βούλησης της Μολδαβίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και θέμα ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να μην μιλήσουμε για τις οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις. Όλοι γνωρίζουμε τις δράσεις της Ρωσίας. Μας ε, την εξήγησαν και καλεσμένοι, γιατί εξασφαλίσε απόλυτο έλεγχο των ΜΜΕ στη Μολδαβία και ο υβριδικός πόλεμος είναι επινόηση της Ρωσίας μέσω και τέτοιων μεθόδων. Και θα πρέπει και εμείς να απαντήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη Μολδαβία ή στην Ουκρανία, αλλά και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια πολιτική παραπληροφόρησης, ε, υπονόμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθούν να δηλητηριάσουν την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και μάλιστα και στις χώρες που έχουν ε, ιδιαίτερα συμφέροντα για τα πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες αλλά και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης προσπαθούν με κάθε τρόπο να σαμποτάρουν τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Ρώσοι. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πώς να αντιδράσουμε. Γιατί σε τελική ανάλυση θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και η Ρουμανία που γειτονεύει με τη δημοκρατία της Μολδαβίας και με την οποία έχουμε και πολλούς κοινού δεσμούς και κοινή ιστορία, και εμείς διαπράξαμε σφάλματα. Προσφέραμε χρήματα στην κυβέρνηση της Μολδαβίας ε, και εφοδιάσαμε ή τροφοδοτήσαμε τον ε, κρατικό προϋπολογισμό της Μολδαβίας χωρίς να γνωρίζουμε πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα θα πρέπει να τα δώσουμε απευθεία στο λαό της Μολδαβίας, στους Μολδαβούς. Γιατί θα πρέπει να κερδίσουμε τις καρδιές και τα μυαλά των Μολδαβών. Γιατί το ίδιο συμβαίνει στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στον κόσμο και στις χώρες Βαλτικής. Γιατί αν ο λαός της Μολδαβίας αντιληφθεί ότι η καθημερινότητά του θα βελτιωθεί και η ευημερία θα αυξηθεί αν στραφούν προς τη Δύση, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα κερδίσουμε αυτή τη χώρα ε, υπέρ των ευρωπαϊκών αξιών της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της οικονομίας αγοράς, υπέρ του κράτους δικαίου, του, της διάκρισης των εξουσιών και ούτω καθεξής. Έτσι θα τους προσετεριστούμε. Αυτές τις αξίες θα πρέπει να προωθήσουμε, όχι μόνο στη Μολδαβία, αλλά παντού. Τι κάνουμε για να αντικρούσουμε τη Ρωσία. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ρωσία επιδιώκει την ε, ικανοποίηση των δικών της συμφερόντων. Ποια είναι όμως τα συμφέροντα Τη Ευρωπαϊκή Ένωση, των ευρωπαϊκών χωρών. Ποια είναι τα συμφέροντά μα, ακόμη και για τη Μολδαβία. Θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ε, στου Μολδαβού, ότι θα πρέπει να έρθουν μαζί μα. και ενδεχομένω να ενταχθούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η θέση του είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με του υπόλοιπου Ευρωπαίου και όχι στον Ευρωασιακό χώρο. Δεν έχουν καμία σχέση με την Ασία οι Μολδαβοί. Επίσης η γλώσσα τους είναι λατινογενής είναι Λατίνοι η Μολδαβοί. Δυστυχώς επί Σοβιετική Ένωσης η Ρωσία υπονόμευσε την ε, κατάσταση στη Μολδαβία και πολλοί και Μολδαβοί και Ουκρανοί και άλλες ε, και άλλοι από τη Σοβιετική Ένωση μετήκησαν προς τη Μολδαβία και μάλιστα τους δόθηκαν και κίνητρα για να μετακομίσουν τη Μολδαβία και να τροποποιήσουν τη δημογραφική της σύνθεση και την ε, να ενισχύσουν την παρουσία των ρωσόφωνων εκεί. Ακόμη και στις αρχές του 20ου αιώνα, οι Μολδαβοί ζούσαν σε αυτή την απομακρυσμένη περιοχή, ε, πολύ περισσότεροι από ό,τι σήμερα, σε ολόκληρη τη Μολδαβία. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε την πολιτική μας συνδρομή και αρρωγή προς τη Μολδαβία και το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και για την Ουκρανία, γιατί φαίνεται ότι και εκεί κάνουμε λάθη στην Ουκρανία. Γιατί δεν τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την ε, Ουκρανία. Έτσι ρίχνουμε νερό στο μήλο της Ρωσίας και της δίνουμε εφόδια να μας πολεμήσει. Θα πρέπει να δώσουμε προπτική στη Μολδαβία και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των Μολδαβών. Γιατί στηρίζουμε πολλές χώρες, βοηθάμε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε περισσότερο και το λαό της Μολδαβίας, να, να δίνουμε περισσότερες υποτροφίες σε Μολδαβούς πολίτες. Να ενθαρρύνουμε τους Μολδαβούς να αισθανιστούν τις αξίες μας. Γιατί στη τελική ανάλυση μιλάμε για κοινέ αξίες σε ένα χώρο ειρήνης, σταθερότητας, ασφάλειας και για το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Σας ευχαριστώ, λυπάμαι, αλλά περιμένω στις 10 μία ομάδα επισκεπτών γιατί θα συναντήσουμε κάποιον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει να φύγω. Πολύ θα ήθελα να παραμείνω εδώ με τους φίλους και αδερφούς από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Σας ευχαριστώ. Έχουμε ως συνήθως ε, κάλυψη web streaming, οπότε μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση. Ο κύριος Οστρεβίτσιος, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους σας για τις παρουσιάσεις τους. Πρέπει να αποφύγουμε την μονομερή περιγραφή της όλης κατάστασης δεν είναι ότι με μία κίνηση τώρα στις 10 η ώρα θα ψηφίσουμε στήριξη προς τη Μολδαβία. Όλα εξαρτώνται από τους πόρους, δηλαδή σύμφωνα με την περιγραφή αυτή, ότι θα δοθούν λεφτά και επομένως θα, σω... θα σωθεί η Μολδαβία. Είναι λανθασμένη αυτή η περιγραφή. Δείτε την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την τοποθέτησή της σχετικά με την ε, στήριξη την οικονομική. Εάν το δούμε καθαρά οικονομικά, τότε είμαστε καταδικασμένοι. Απλώς βασιζόμαστε σε κάποια μακρομεγέθη οικονομικά, τα οποία στην πραγματικότητα δεν μας λένε τίποτα. Η νόσος, επί της οποίας έχετε το δίκιο, δηλαδή η εξαφάνιση της αντικειμενικής κανονικής λέει ο δημοσιογραφία στη Μολδαβία ξεκίνησε πριν από πάρα πάρα πολύ καιρό. με την μεταστροφή της αγοράς των μέσων σε μονοπόλιο, την κατάργηση της ελευθερίας του τύπου, γιατί λυπάμαι και για αυτό πρέπει να μιλήσουμε, καμία αντικειμενικότητα, μία περιγραφή των πραγμάτων που δεν αποτυπώνει τα πράγματα παρά μόνο ασπρόμαυρα, ας το πούμε, και δεν δίνει την αληθινή του διάσταση. Και αν βασιστούμε λοιπόν σε κάποιες λανθασμένες παραμέτρους της περιγραφής, δεν θα καταλάβουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τους ε, πολιτικούς εκπροσώπους Μολδαβίας εξαρτάται και από τη δική μας τάση. Υποτίθεται ότι πρέπει να υποστηρίζουμε τα πολιτικά κόμματα που τοποθετούνται φιλικά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια καθημερινή διαδικασία υλοποίησης της όλης σχέσης σύνδεσης. Και όσο περισσότερο υλοποιείται το θεματολόγιο της σύνδεσης, τόσο περισσότερο μπαίνουμε στο έλος, στην κινούμενη άμμο που είναι η κατάσταση της Μολδαβίας. Πρέπει λοιπόν να μην υπεραπλωστεύουμε προνατοικούς, αντινατοικούς κτλ. Το μολδαβικό έθνος και ας το αποκαλέσουμε όπως ονομάζεται, πλησίασε και απομακρύνθηκε από τη ρωσοποίηση σε ένα ελεγχόμενο κοινωνικό περιβάλλον. Πρέπει να είμαστε απολύτως ανοιχτοί και απολύτως ειλικρινείς στην περιγραφή μας και στην ανάλυση μας. Και μεταξύ των αξιών και του οικονομικού συμφέροντος και της διαπλοκής τους κάποιων πολιτικών που τοποθετούνταν για αυτά τα πράγματα με κομψό τρόπο, δεν βλέπω καμία επίλυση εάν δεν καταφέρουμε να κατανοήσουμε πρώτα απ' όλα σωστά την κατάσταση. Έχουμε σημαντική και πραγματική παραπληροφόρηση. Και έχουμε μια διαδικασία με βασικές κατευθύνσεις που οδηγούν σε μια τυφλή κοινωνία. Δεν θέλω να επικρίνω καμία πολιτική δύναμη. Αλλά κανείς μπορεί να χειρίζεται τα πράγματα με το δεξί του χέρι ή το αριστερό του χέρι, λέει ο μιλτής. Στην πραγματικότητα πρέπει να κινείται κανείς ε, με διαδικασίες από κάτω προς τα πάνω, με συμμετοχικότητα, ώστε η πραγματική ερευνητική δημοσιογραφία να επανέλθει στο προσκήνιο στη Μολδαβία και να αποτυπώνει τα πράγματα όπως είναι. Ήθελα να μας πείτε λίγο περισσότερα για τον κρατικό φορέα της τηλεόρασης, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω υποστηρίζεται πληρέστατα ε, οικονομικά Έχουμε κάποια μέσα ενδυνάμωσης των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης που προτείνονται. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάποια περισσότερα πράγματα για τη θέση που έχει λάβει το Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Οι πολιτικοί εκπρόσωποι πώς τοποθετούνται όταν κοιτούν την κατάσταση της χώρας Δηλαδή μια μακροοικονομική επέμβαση, διάσωση θα είναι επαρκής αν δεν λάβουμε άλλα μέτρα που νομίζω ότι είναι απαραίτητα και εγκαίρως. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σαφχάουζα. Κοιτάξτε, καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Στρεβίτσιους και να τον συγχαρώ. Εδώ έχουμε απέναντί μας, Πρόεδρε, ένα περίπλοκο παιχνίδι. Ο κύριος Ντοντών που υπήρξε κομμουνιστής και τώρα προβάλλει τις χριστιανικές αξίες. Ε, ο Παβέλ Φιλίπ ε, που είναι συνδεδεμένος με συμφέροντα ολιγαρχών έχουμε απέναντί μας ένα πολύ περίπλοκο, πάρα πολύ περίπλοκο πολιτικό σκηνικό, σύστημα, παιχνίδι που δεν μπορούμε απλώς να το αναλύσουμε στους φιλοευρωπαίους ή αντιευρωπαίους, φιλορώσους ή αντιρώσους γιατί έχουμε συνδέσμους πολλών επιπέδων και περίπλοκους προς όλες κατευθύνσεις. Ας μην υπεραπλουστεύουμε λοιπόν και με την επιλογή των ε, ομιλητών μας. Μιλούμε για μια χώρα που βρίσκεται σε ένα στρατηγικό σημείο γεωπολιτικά μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε γέφυρες, να βρούμε διόδους, να βρούμε ε, τρόπους συμφιλίωσης σε ένα κοινό έργο, σε μια κοινή κατεύθυνση και ας μην τοποθετούμε την ε- Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της στο ένα ή στο άλλο στρατόπεδο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ρωσία είναι δύο κόμβοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας άλλος ανεξάρτητος. Και μιλούμε λοιπόν για μια χώρα που τοποθετείται σε ένα κρίσιμο επαναλαμβάνω γεωπολιτικό σημείο και πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες ιδιαίτερα που σχετίζονται με τα μέσα ενημέρωσης. Θυμίζω ότι ολόκληρο το σύστημα μέσων ενημέρωσης ήταν κατά του Τραμπ στην Αμερική. Ολόκληρο το σύστημα ενημέρωσης στη Γαλλία είναι κατά της Λοπέν και δεν μας εμφανίζουν ως χώρα πρότυπο ως προς τα μέσα ενημέρωσης. Τα μέσα ενημέρωσης τάσσονται με το mainstream τα βλέπουμε αυτά πολύ συχνά και πρέπει κανείς να τα επικρίνει και να τα αντιμετωπίζει αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, δεν είναι τόσο άσπρα και μαύρα. Ενέχονται πάρα, πολλές, πάρα πολλά επίπεδα κοινωνιολογικής ανάλυσης, αν θέλετε να το πούμε έτσι, και πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τους σπόρους που προσφέρουμε. Από τα τέσσερα δισεκατομμύρια, τα δύο δεν ξέρουμε που κατέληξαν πρέπει να το ελέγξουμε κάπως και θα συμφωνούσα απολύτως ε, με τον συνάδελφο που μόλις ε, απεχώρησε ότι πρέπει να ενισχύουμε όχι τον προϋπολογισμό γενικά αλλά συγκεκριμένα έργα και μόνο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και την εικόνα και την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνολική δηλαδή ευρωπαϊκή πολιτική που πρέπει να στρέφεται όλο και περισσότερο προς τους πολίτες και όχι σε ένα κεντρικό επίπεδο. Ο ρόλος μας δεν είναι να υποστηρίξουμε, να υποδαβλήσουμε μια αντιπαράθεση μεταξύ των φίλων ή αντιευρωπαίων, αλλά να βοηθήσουμε την κοινωνία συνολό τη. Σας ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κέλαμ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσθέσω σε αυτά που είπαν εκεί οι προηγούμενοι μιλητέ, ότι οι καταστάσεις είναι σχετικά απλές κάποιες φορές. Και όταν το παρουσιάζουμε αυτό ως περίπλοκο, είναι ουσιαστικά μια απόπειρα να αποφύγουμε την πραγματικότητα, την αλήθεια, να την κοιτάξουμε ακατάματα. Και μιλάω για τη ρωσική επιρροή. Ξέρουμε ότι τα ρωσικά χρήματα πηγαίνουν στην εξαρτία της κυρίας Λεπέν εδώ και χρόνια. Πρόεδρε, πρόεδρε. Και ένας από τους ε, διαμεσολαβητές είναι και εδώ στην αίθουσα. Με εντυπωσίασε ιδιαίτερα πάντως ε, η παρουσίασή σας, ε, κυρία Μωράρη και κύριε Μάκοβέη. Εγώ επί δεκάδες χρόνια ε, έζησα στην υποσυγκριτική κατοχή Εσθονία και αντιμετώπισα την πρόκληση της του μονοπωλίου πληροφοριών και της παραπλάνησης. Αλλά τότε ήταν απλά τα πράγματα. ήταν απλό να ξέρουμε πότε ακούμε προπαγάνδα. Τώρα νομίζω ότι μπορεί να αισθάνεται κανείς ανεξάρτητος, αλλά παρόλα αυτά να περιτριγυρίζεται από αόρατα τείχη παραπλανητικών πληροφοριών και ακόμα ο κόσμος είναι φλακισμένος στο παρελθόν του. Υποστηρίζω πραγματικά τις ιδέες. Την ιδέα μάλλον ότι και η Μολδαβία θα πρέπει να διαλέξει και να επιλέξει είτε την ε, σύγχρονη Ευρώπη είτε το σοβιετικό παρελθόν. Είναι δύσκολη η επιλογή, αλλά το μήνυμά σας είναι σημαντικό. Γιατί δεν ακούμε, θεωρώ και δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο είναι να γίνει μια αλλαγή στο κεφάλι του κόσμου στην οτροπία του κόσμου και πόσο πολυσύνθετη και έντεχνη είναι αυτή η προπαγάνδα βρώμικες επιχειρήσεις, οικονομικά συμφέροντα, διαφθορά. Και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε σε πρώτη φάση είναι να δώσουμε μια σαφή ευρωπαϊκή προοπτική στη Μολδαβία. Γιατί διστάζουμε και αν φυτελαντευόμαστε. Θα πρέπει να στείλουμε ένα σαφέ μήνυμα ότι είναι δικαίωμα τη Ευρωπαϊκή Μολδαβία να ανήκει στη... και να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. η κυρία βάση του δικού μα μήνυματο. Σα φυσικά. Αυτή θα πρέπει να είναι η κύρια βάση του δικού μα μηνυματο σα θέλουμε. σα θέλουμε σε κάποια χρόνια στου κολπου τη ενωση Το θέμα είναι το πώς θα υποστηρίξουμε πραγματικά τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωση και η κυρία Κίφερ το ανέφερε. Υπάρχει το Euronews στη ρουμανική γλώσσα στον κόσμο στη Μολδαβία. Διατίθεται. Όχι. Σχόλια εκτός Τι γίνεται με τις ε, διαδικτυακές επικοινωνίες. Και ποια είναι η στάση, η προσέγγιση στο σοβιετικό παρελθόν, στην πρόσφατη ιστορία της Μολδαβίας δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό. Ξέρουμε όλοι ότι όλες οι σοβιετικές χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό, το πώς θα αντιμετωπίσουν την πρόσφατη ιστορία τους, πώς θα την χειριστούν πώ θα χειριστούν αυτό το αυταρχικό καθεστώ του παρελθόντο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, με πάρα κύριε Κέλαμ, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τελευταίο αυτό τμήμα κυρίω τη παρέμβασή σα, με το οποίο συμφωνώ όλο ιδιαίτερου. Ο κύριος Μπορτινάρου, πριν πάρετε το λόγο να σας ενημερώσω κύριε Σαφχάουζερ, ότι έχετε μισό λεπτό at bottom. Να προετοιμαστείτε προσεκτικά, γιατί θα σας διακόψω στα 30 δευτερόλεπτα, δεν έχουμε χρόνο. Ο κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μισό λεπτό για μένα μετά. Ναι. Προς ε, έκπληξη πολλών συναδέλφων και των ε, ε, επωνομεζόμενων εμπειρογνωμόνων θα μιλήσω την ίδια γλώσσα με τον κύριο Μακοβέη μιλάω την ίδια γλώσσα με τον ε, κύριο Μακοβέη και δεν είναι αυτό ισχυρή απόδειξη ότι η ρουμανική και η μολδαβική γλώσσα είναι σχεδόν ταυτόσιμες. Εν πάση περιπτώσει, αφήσουμε αυτό το ζήτημα. Όλα αυτά που ακούσαμε και μας παρουσιάστηκαν επιβεβαιώνουν αυτά που ξέραμε ή τέλος πάντων τα οποία θεωρούσαμε δεδομένα. Η Μολδαβία και τα άλλα κράτη τα οποία ανήκαν στη Σοβιετική επιρροή αποτελούν θέατρο βίαιων στρατηγικών συγκρούσεων. Το ίδιο έγιναν και στην Γεωργία, στη Μονταβία, στην Ουκρανία και σχεδόν παντού. Όχι επειδή είναι από τη φύση της επιθετική η Δύση, αλλά επειδή η Ρωσία του Πούτιν θέλει να δημορφώσει εκ νέου αυτή τη σφαίρα επιρροή τη. Είναι ένα υβριδικό, ε, είναι ένα υβριδικό πόλεμο. Αυτό ίσω είναι ο πιο σωστό ορισμό ε, στην προκειμένη περίπτωση. Το πιο γνωστό καφενείο, ξέρετε, είναι, έχει την επωνυμία προπαγάνδα. Τυχαίο. Αυτό νομίζω ε, ότι καταδεικνύει και τις σχέσεις με τη Ρωσία. Δύο ερωτήσεις λοιπόν θα ήθελα να σας θέσω για τη μου και κάτι άλλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε, μάλλον τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να υποστηρίξει και να βοηθήσει τις χώρες αυτές της Ανατολικής Γειτονίας και προκειμένου να φροντίσει κάτι να μπορέσουμε να κάνουμε κατά της διαβρωτικής αυτής επιθετικής προπαγάνδας, όχι μόνο στη Μολδαβία αλλά και στις άλλες ε, χώρες και να σας πω και το εξή στις ε, Ηνωμένες Πολιτείες, στην Γαλλία, στη Γερμανία. Όταν εκεί υπάρχουν ανησυχίες ε, για την επιρροή από τη Ρωσία, για τους μηχανισμούς μέσω των οποίων ε, ενδεχομένως επεμβαίνει η Ρωσία. Αν εκεί υπάρχουν ανησυχίες, φανταστείτε πόσο ευάλωτες είναι αυτές οι προσβητικές δημοκρατίες στη ρωσική προπαγάνδα. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε σε ό,τι αφορά αυτά τα πάκετα υποστήριξη. Αναρωτιέμαι κατά πόσον θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τα κρατή αυτά να αναπτύξουν και δικές τους ικανότητες, δικές τους ε, μηχανισμούς για την καταπολέμηση της προπαγάνδας σε αυτόν τον ευρετικό πόλεμο. Γιατί αν ε, κερδίσουν τον πόλεμο σε αυτό το χώρο, Ποιο θα είναι ο επόμενο χώρο όπου θα δοθεί ο πόλεμο τη προπαγάνδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ασταθή χώρο, ξέρετε, και νομίζω ότι τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν αυτό εν μέρη. Αυτό ο αγώνα στον τομέα τη ενημέρωση, αυτό ο πόλεμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει όντω συγκεκριμένη άρρωγη προ τι χώρε αυτέ. Το συνταγματικό δικαστήριο της ε, Μολδαβικής Δημοκρατίας αποφάνθηκε ότι η Μολδαβία, μάλλον η υπερνιστερία αποτελεί ουδέτερο κράτος και υπάρχει δυνατότητα και το δικαίωμα να κλείσει στρατιωτικές συμμαχίες για την προστασία της. Ε, αυτό είναι κάτι το πολύ τολμηρό και θα πρέπει να υποστηριχθεί. Κύριε Μποστινάρου, λέει η Πρόεδρος. υπήρξε κάποια παρανόηση σε αυτά που είπατε. Σας παρακαλώ, για πείστε ξανά αν θέλετε αυτό το κομμάτι για την υπερμυστερία, γιατί γνωρίζω πώς έχει η κατάσταση. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι βεβαίως, λέει ο κ. Μποστινάρου. Προχθές το Στοχματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας αποφάσισε, αποφάνθηκε ότι η χώρα ε, ενώ αποτελεί ουδέτερο κράτος, έχει το δικαίωμα να προσχωρήσει σε μια στρατιωτική συμμαχία προκειμένου να προασπίσει την ενταφική της ακαιρεότητα και την επικυριαρχία της σε ό,τι αφορά κατοχή ή υπερδνηστερία, η υπερδυνεστερια η θεωρείται από το Διεθνές Δίκαιο ως κατεχόμενο τμήμα ενός επικυριαρχού κράτους. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το, το συνταγματικό δικαστήριο λοιπόν αποφάσισε να αποφανθεί ούτω. Τώρα. Στι τελευταίε δύο εβδομάδε, ο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατία τη Μολδαβίας αποφάσισε να συνεργαστεί θεσμικά με το FBI για να καταπολεμήσει, να αντιμετωπίσει ε, το, τη μάστιγα του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς σε υψηλά πολιτικά κλιμάκια και γνωρίζοντας ότι οι ικανότητες της Μολδαβίας είναι πολύ περιορισμένες στον τομέα αυτό και επειδή έχουν να αντιμετωπίσουν ε, το τεράστιο κύκλωμα της διαφθοράς που ένα τμήμα του έχει ε, διασυνδέσεις με ρωσικές ε, εγκληματικές οργανώσεις και συμμορίες και όχι μόνο με ρωσικές συμμορίες Πάντως είναι πολύ ψηλό το επίπεδο διασύνδεσης. Εξού και η έκκλησή μου προς τους συναδέλφους. Πριν να αποφασίσουμε ε, την σύνδεση με το ΕΛΚ, ε, ε σημαίνει ότι είναι ε, καλό ε, φιλοευρωπαϊκό, ενώ αν ε, συνδεθεί με, το, με τους σοσιαλιστές είναι κακό. Θα πρέπει να δούμε τι κάνουν, τι κάνει η κυβέρνηση. Να δούμε το γενικότερο πλαίσιο. Δεν είναι όλα μαυρά-άσπρα, υπάρχουν και άλλες αποχρώσεις. Ούτε είναι μόνο μαύρα ή μόνο άσπρα. Θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες, τις αποχρώσεις, να εξασφαλίσουμε την επιβίωση της χώρας και να παραμείνει ζωντανή η, ο δυτικό προσανατολισμός και όχι μόνο σε επίπεδο διακηρύξεων αλλά και εμπράκτος και να αξιολογήσουμε κάθε δέσμη μέτρων αρρωγής ε, ε, με βάση τα αποτελέσματα που προσφέρει η κυβέρνηση. Μόνο έτσι θα φύγει η χώρα από το διέξοδο. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε φακούς των Βρυξελών και να χαρακτηρίζουμε κάτι μόνο καλό ή μόνο κακό. Έτσι θα χάσουμε αυτή τη χώρα, θα την προσφέρουμε ε, και δωρεάν μάλιστα στο πιάτο στη Ρωσία με μια τέτοια συμπεριφορά. Ε, κύριε Σαφχόζερ, παρακαλώ τηρήστε το μισό λεπτό που σας έδωσα γιατί θα πρέπει να ακούσουμε και τους καλεσμένους μας. Έχω και εγώ κάποια σχόλια μετά από σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ καταρχήν που μου δίνετε έστω και μισό λεπτό. Θα ήθελα απλώς να πω στον συνάδελφο Κέλα ότι δεν θα μου δώσετε εσεί μαθήματα για την καταπολέμηση του κομμουνισμού. Εγώ έδωσα ε, μάχη, αγωνίστηκα κατά το, του κομμουνισμού, πολύ πιο έντονα από ότι εσεί, κύριε Κέλαμ. Σε ό,τι αφορά ε, τις μου με τη Ρωσία από το 1992, ε, όταν ήμουν στο Συνταγματικό Συμβούλιο και το 1995, όταν στην πρώτη επίσκεψη του Σιράκα έγραψα άρθρο για να προωθήσω αυτή την ε, συνεργασία. Δεν... Ε, δεν ε, είναι πρόσφατη σχέση μου με τη Ρωσία, ούτε ανάγονται στην συμμετοχή μου στο εθνικό μέτωπο. Βλέπετε πολύ κοντόφθαλμα τα πράγματα και στο επίπεδο της δικής σας ποταπότητας τα αντιμετωπίζετε όλα. Ευχαριστώ. Μην αρχίζετε τώρα προσωπικές συζητήσεις ε, ad hoc. Παρακαλώ, παρακαλώ συνάδελφοι. Συμφωνώ και με τον κύριο Στρεβιτσίους ε, και με άλλους ομιλητές ότι διαπιστώνουμε πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση μετά τις παρουσιάσεις και των καλεσμένων μας ε, και σε πολιτικό επίπεδο. Και σίγουρα δεν είναι δεν θα πρέπει να είμαστε μονόπλευροι, να υπεραπλουστεύουμε τα πράγματα. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες κατευθυντήρες γραμμές που καλό θα ήταν να ακολουθήσουμε. ώστε να ξεκινήσουμε αυτό το δρόμο της αξιολόγησης ε, της κατάστασης στη Μολδαβία, ώστε να εφαρμόσουμε τις σωστές και κατάλληλες λύσεις. Και αυτό προϋποθέτει μια αξιολόγηση των τρόπων του, της προπαγάνδας που γίνεται αυτή τη στιγμή, αυτού του επικοινωνιακού πολέμου που λαμβάνει η χώρα στη Μολδαβία. Και μετά τις παρεμβάσεις και των συναδέλφων. Αποκόμισα την, την εντύπωση, λαμβάνοντας υπόψη και τα σχόλια του κυρίου Κέλαμ για την ανάγκη να ε, ξεκαθαρίσει η θέση της κοινωνίας απέναντι στο σοβιετικό παρελθόν. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και του δικού μας κόσμου, γιατί ένα τίμα αφορά την ξεκαθάριση, το ξεκαθάρισμα με το σοβιετικό παρελθόν. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι να αντιληφθούμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι πολλές κοινωνίες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης είναι αρκετά παραδοσιακές και δυστυχώς ο Πούτιν κατάφερε να προβληθεί και στις κοινωνίες της Ευρώπης ως ε, αμύντορας των παραδοσιακών αξιών, ως προστάτης των παραδόσεων. Και αυτό πραγματικά είναι ε, τραγική ηρωνία ε, της πολιτικής να επιτρέψουμε σε έναν πρώην συνταγματάρχη της ΚΑΚΕΜΠΕ να προβάλλεται ως ε, προασπιστής ε, των ε, παραδοσιακών αξιών. Και γνωρίζοντας την ιστορία και γνωρίζοντας τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από μια τέτοια οργάνωση, είναι πραγματικά το άκρο των αλλά είναι γνωστά αυτά από ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου. Οπότε δεν υπάρχει καμία α, ταύτιση της Ρωσίας με τις παραδοσιακές αξίες, ούτε υπάρχει καμία εξίσωση ή ταύτιση της Ρωσίας και της σλαβικής προέλευσης. Και οι Πολωνοί είμαστε Σλάβοι. 100%. Απολύτως. Αλλά ε, όχι μόνο ο Πούτιν, οι Ρώσοι γενικώ προσπάθησαν να μεταλαμπαδεύσουν αυτή την εσφαλμένη εντύπωση, η ιδέα ότι όλοι οι Σλάβοι είναι Ρώσοι, ότι η Ρωσία και Ρώσοι και Σλάβοι ταυτίζονται. Αυτό το όμως μια υπεριλιστική τακτική. Είχαμε 123 χρόνια του διαμελισμού της ε, Πολωνίας και της υποταγής της Πολωνίας στη Τζαρική Ρωσία και στη κατοχή από τη Τζαρική Ρωσία. Είχαμε πολλές εξεγέρσεις των Πολωνών και όλοι στην προσωπική του ιστορία είχαν πολλά χρόνια αγώνα κατά της Ρωσίας και μας μεταχειρίστηκαν ως Σλάβους προδότες έτσι μα φέρθηκαν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι Ρώσοι έχουν το προνόμιο ή το δικαίωμα να εκπροσωπούν όλους τους σλαβικού λαούς, όλα τα σλαβικά έθνη. Και δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε Ευρωπαίοι επειδή δεν είμαστε Σλάβοι. Γιατί κάτι τέτοιο προσπαθούν να προβάλλουν. Γι' αυτό περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Φυσικά το αντιλαμβάνομαι και έχετε δίκιο ότι η προέλευση, η γλώσσα, ο πολιτισμός, η κουλτούρα ε, είναι κάτι κοινό και ε, ένα κοινό μας στοιχείο είναι ότι ανήκουμε σε αυτή την λατινική κουλτούρα, όχι μόνο λόγω της γλώσσας, αλλά είμαστε και τη μέτα της Ρωμακαθολικής Εκκλησίας. Και αυτό είναι ο κοινό ε, παρανομαστής ε, της καθολικής Εκκλησίας, αυτό το λατινικό παρελθόν. Θα πρέπει πάντως να βρούμε τα σωστά μέσα για να αντιμετωπίσουμε και αυτό το θέμα των χριστιανικών αξιών. Για να αγγίξουμε τους πιστούς που θέλουν να παραμείνουν ορθόδοξοι και εντός της Μολδαβίας και που έχουν κάθε δικαίωμα να ανήκουν στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, στην ευρωπαϊκή κουλτούρα. Επίσης, παρουσιάζοντας μια θετική εικόνα μας στη Μολδαβία, θα πρέπει να βρούμε και ένα μήνυμα προς αυτή την ομάδα του πληθυσμού. Δεν σημαίνει ότι οι χριστιανοί ορθόδοξοι είναι πιο κοντά στη Ρωσία. Άλλωστε, οι δεσμοί είναι μάλλον δεσμοί υποταγής των Ορθόδοξων εκκλησιών στην Ευρώπη. Και αυτό καθιστά ακόμη πιο περίπλοκη την κατάσταση. Οπότε δεν θα πρέπει μόνο να ε, επισημάνουμε το έργο και το ρόλο της ε, Εκκλησίας ε, και να βρούμε και ένα θετικό μήνυμα για να αποδεσμεύσουμε την Εκκλησία και να βρούμε ένα θετικό μήνυμα προς τους ε, Μολδαβούς, προς Ευρωπαίους και άλλους που θέλουν να παραμείνουν ταυτόχρονα και χριστιανοί, ορθόδοξοι και Ευρωπαίοι. Γιατί είναι δύσκολο να κάνουμε μια σαφή τομή μεταξύ της Ασίας και της Ευρώπης. Η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή άσπρο-μαύρο, είναι πιο πολυσύνθετη. Και στην ε, έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Stratcom το επισημάναμε. Βέβαια ήταν πολύ ακροθυγής αυτή η μία για τις ε, εκκλησίες, αλλά θα πρέπει να βρούμε ένα θετικό αφήγημα και για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Τώρα θα ξαναδώσω το λόγο στους καλεσμένους μας και γιατί ο χρόνος δυστυχώς είναι πολύ περιορισμένος με την ίδια σειρά που μίλησαν και προηγουμένως. Περισσότερο ακούσαμε παρατηρήσεις παρά απορίες, οπότε είναι πιο εύκολο και για σας. Είπα με την ίδια σειρά που μιλήσατε και προηγουμένως. Πρώτα κυρία Κίφερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το σχόλιο του κυρίου Κίλαμ σχετικά με το 48% μέσω της ε, προεκλογικής εκστρατείας ε, που επετεύχθη μέσω διαδικτυακής προσπάθειας. Νομίζω ότι μέσω του ίντερνετ, μέσω του διαδικτύου ε, μπόρεσε να πλησιάσει σε ένα κοινό ένα κοινό που τοποθετείται πιο φιλοευρωπαϊκά θα μπορούσαμε να, να το πούμε έτσι και την ίδια δίωδο προσπαθούμε και εμείς να χρησιμοποιήσουμε. Ο κύριος Σιγκάλε αναφέρθηκε στη συνεργασία Έχουμε συναδέλφους από πολλά κράτη-μέλη που έχουν και τα δικά τους δίκτυα στις ε, πρωτεύουσε. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε όλη αυτή τη δικτύωση εν ζωή. Αυτός ο συντονισμός βεβαίως θα μπορούσε να ενισχυθεί Μερικές φορές ε, την πληροφορία την κατέχουν κρατικοί φορείς οι οποίοι δεν έχουν ιδιαίτερη διάθεση να μοιραστούν την πληροφορία αυτή, αλλά είναι και θέμα πολιτικής βούλησης. Ο κύριος ε, Μπουστινάρου ε, ρώτησε τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την προπαγάνδα αυτή. Είναι πολύ σαφές από τις τοποθετήσεις των δύο προσκεκλημένων ότι τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης χρειάζονται τη βοήθειά μας και είναι ε, θετικό που βλέπουμε ότι η Κομισιόν έχει την πρόθεση να ενισχύσει και καλό θα ήταν να μην μιλούμε μόνο για προγράμματα κατάρτισης και ο κ. Μακοβέη θα μπορούσε να το επιβεβαιώσει. Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι το τρέχον κόστος για να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις αυτές των μέσων ενημέρωσης. Αλλά αν σας ενδιαφέρει το θέμα θα σας ενθάρρυνα να κάνετε μια τέτοια συζήτηση, ένα τέτοιο διάλογο για να καταλάβετε καλύτερα τα επίπεδα του θέματος και πρέπει να ενισχύσουμε όλη την προσπάθεια στρατηγικής ενημέρωσης και επικοινωνίας προκειμένου όμως να επιτύχουμε τη θέμενη αξία ε, χρειαζόμαστε ανθρώπινους πόρους, χρειαζόμαστε ειδικευμένους ανθρώπους στις ευρωπαϊκές αποστολές για να δαπανώνται αυτοί οι πόροι αποτελεσματικά και σωστά. Αυτή τη στιγμή οι δαπάνες αυτές δεν γίνονται με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Στρεβίτσιους. Είναι και πολιτική η προσπάθεια που θα μπορούσαμε να καταβάλουμε. ώστε να αντιμετωπίσουμε την διαφθορά και βεβαίως κάτι που δεν είναι επίσημη θέση της υπηρεσίας μας δίνοντας μακροοικονομική βοήθεια δεν θα είναι θετικό το αποτέλεσμα για την φήμη, για την εικόνα μας. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Μωράρια. I have some small Κοιτάξτε, για την επιρροή του διαδικτύου, τα καλά νέα είναι τα τελευταία δύο χρόνια οι χρήστες του ίντερνετ αυξάνονται μαζικά. Έχουμε ήδη μια γενιά που δεν παρακολουθεί τηλεόραση, αυτό είναι καλό, αλλά έχουμε ακόμα το 80% του συνολικού πληθυσμού που χρησιμοποιούν ως πρώτη πηγή ενημέρωσης την τηλεόραση. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ελπίζω ότι σε πέντε χρόνια η κατάσταση θα είναι καλύτερα, αλλά μέσα σε αυτά τα πέντε χρόνια θα έχουμε δύο εκλογές. Και τι θα συμβεί με την τηλεόραση να παραμένει πρώτη πηγή ενημέρωση. Ο κύριος Γκάλε αναφέρθηκε σε κάποιες προϋποθέσεις στήριξης. Μα μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε την Μολδαβία, διότι τα τελευταία 7 χρόνια από το 9 είχαμε μια απολύτως ανοιχτή διάθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια άμεσες ενισχύσεις από Ευρωπαίους δωρητές και είναι πολύ σημαντικό αλλά ξέρετε τι συνέβη με αυτά τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν με απολύτως αδιαφανή τρόπο έγιναν κάποια θετικά πράγματα αλλά τροφοδότησαν τις μεγαλύτερες υποθέσεις διαφθοράς στην ιστορία μας, τη σύντομη ιστορία μας. Όλη αυτή λοιπόν ότι η ευρωπαϊκή στήριξη αυτή συνεδέθη με διαφθορά υψηλού επίπεδου. Με πρώην Πρωθυπουργό που είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή, με ξέπλυμα χρήματος στο μολδαβικό τραπεζικό σύστημα. Επομένως βεβαίως και χρειάζονται αιρέσεις και προϋποθέσεις δεν είναι μόνο η ρωσική προπαγάνδα αλλά και μια πολύ διεφθαρμένη ελίτ του πολιτικού συστήματος και αυτή πολύ συχνά δεν επεκρίθη από τους Ευρωπαίους εταίρους. Πολύ συχνά όταν έπρεπε να αναφερθούν σε περιπτώσεις σκανδαλώδης διαφθοράς δεν το έπραξαν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί. Και πολύ συχνά στο κοινό περνάει η εικόνα ότι με αυτόν τον τρόπο, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει διαφθαρμένους πολιτικούς, είναι και η ίδια διαφθαρμένη. Ο κύριος Στρεβίτσιος, να σας ευχαριστήσω μάλιστα για τη στήριξή σας. Ρωτήσατε με ποιο τρόπο το Κοινοβούλιο της Μολδαβίας αντέδρασε σε όλη αυτή την προπαγάνδα και αν προσπάθησε να κάνει κάτι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 2015 προσπάθησαν επιθετικά σχεδόν να προωθήσουν έναν, μια πράξη νόμου κατά της ε, ε προπαγάνδας από ένα πολιτικό κόμμα συγκεκριμένο διοργανώθηκαν ε, διάλογοι, debate, ζητήσει και δεν έγινε τίποτα. Μόνο το δικό μας κανάλι απομακρύνθηκε από τη ρωσική προπαγάνδα ο, ο, ο κύριος Ποχότνιου δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και τώρα περιμένουμε νέες τροποποιήσεις του ραδιοτηλεοπτικού κώδικα από την αρχή Οκτωβρίου ίσως για να δούμε πώς θα επηρεάσει όλους αυτούς τους σταθμούς γιατί όλοι θα είναι υποχρεωμένοι να έχουν 8% τοπικού περιεχομένου. και θα δούμε αν ο φορέας των τηλεοπτικών μεταδόσεων παρακολουθήσει και ελέγξει όλα αυτά. Μιλάω για την ευρωπαϊκή προοπτική. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αλλά δεν πρόκειται να έχει κανένα αποτέλεσμα χωρί αιρεσιμότητα. Θα χρησιμοποιηθεί απλώ για την εσωτερική προπαγάνδα, για αυτού που επικρίνουν την κυβέρνηση, για την έλλειψη διαφάνεια, για την έλλειψη μεταρρυθμίσεων. Θα ακούμε καθημερινά από του σταθμού του ότι μας επικρίνεται αλλά ε, μας δίνεται απλώς την ευρωπαϊκή προοπτική. Θα κατηγορηθούν δηλαδή ότι είναι πράκτορες των Ρώσων στην ουσία. Σύμφωνα με, ένα, με μια έρευνα του 16, σχεδόν το 60% του πληθυσμού ε, είναι, τοποθετείται ε, με μια θλίψη απέναντι στην κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Και κύριε Μπουστινάρου, ε, μιλήσατε για αυτήν τον... Όταν μιλήσατε για αυτό το καφενείο και την προπαγάνδα, τις συζητήσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών ε, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μία, εγώ είμαι μέλος, την επόμενη συζήτηση θα μιλήσουμε ε, για την ε, θέση των δικαιωμάτων των ομοφιλοφίλων στη χώρα αλλά γίνεται μία προπαγάνδα μέσω του διαδικτύου από την κυβέρνηση κατά των ανθρώπων που κάνουν αντικειμενική και ελεύθερη δημοσιογραφία. Μας επικρίνουν μας κατηγορούν ως πράκτορες των Ρώσων ή οτιδήποτε άλλο, ώστε να απομακρυνθεί το κοινό από εμάς. Ε, ε, επί τρία χρόνια ε, έλεγαν ότι ήμασταν το πιο αντικειμενικό πολιτικό τοξό στην τηλεόραση. Δεν ξέρω αν ένας Ρώσος πράκτορας θα μπορούσε να το έχει καταφέρει. Ο κύριος Μακοβέη, λέει η πρόεδρος, συνάδελφοι, έχουμε πολύ λίγο χρόνο γιατί μετά θα πρέπει να συνεχίσουμε το επόμενο θέμα. Μάλιστα, θα ήθελα να επιβεβαιώσω αυτά που είπε και η συνάδελφό σε ό,τι αφορά για το καφενείο αυτό, για το καφενείο το οποίο ονομάζεται προπαγάνδα και σε ό,τι αφορά την αντικειμενική δημοσιογραφία στην Δημοκρατία τη Μολδαβία. Τα πιο πολλά ζητήματα και ερωτήματα έχουν ήδη απαντηθεί, αλλά να πω και εγώ δύο λόγια. Γιατί θα πρέπει να γίνει εφ' εξή. Θα πρέπει να επενδύσουμε στις ε, εγχώριες, στα εγχώρια ποιοτικά προϊόντα ποιοτικά τονίζω, γιατί τα ρωσικά προϊόντα, ό,τι περνάει και έρχεται από τη Ρωσία, είναι πάρα πολύ δημοφιλές ε, στην ε, Ρωσία. Ε, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια ε, δαπανώνται προκειμένου να υπάρχουν αναλλακτικέ για να υπάρχει ένα καλό μολδαβικό προϊόν για την αλλαγή τώρα των νόμων. Το είπε και η Νατάλια θα εφαρμοστούν αυτά και θα υλοποιηθούν από τον Οκτώβριο. Αλλά θα έχουν αποτελέσματα μόνο αν έχουν και κάποιες δυνατότητες και κάποιες ευκαιρίες η εγχώρη παραγωγή. Και ζητήσαμε λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην προβλέψει μόνο το επόμενο βήμα, αλλά και πιο πολλά βήματα, τα μετέπειτα βήματα στην υποστήριξη της τοπικής παραγωγής, προκειμένου να υπάρχουν πραγματικά καλά και ποιοτικά χώρια προϊόντα τα οποία να τα αντάξουμε στην προπαγάνδα. Κάτι άλλο τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό διαπιστώνοντας ε, ότι και στην αγορά τη διαφήμιση υπάρχει τεράστια μονοπολία και εδώ πέρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί δεν υπάρχει αλλιώ εναλλακτική δυνατότητα σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία του τύπου και των μέσων ενημέρωση. Και η οικονομία καταλαβαίνετε ότι καθορίζει την πολιτική των εκδόσεων και έτσι πάρα πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί, εκπομπές, τηλεοράσεις, σταθμοί ε, ε, πολύ απλά κραχακοπούν γιατί δεν έχουν ε, έσοδα γιατί προφανώ η διαφήμιση ακολουθεί πολλά πολύ γνωστά κριτήρια και υπόκειται σε εσωτερική χειραγώγηση και σε προεκλογικούς αγώνες αλλά προφανώς και σε άλλε κρίσιμε εποχές. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Ευχαριστούμε τον κύριο Μακοβέη. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πειθαρχία που δείξατε σε ό,τι αφορά το χρόνο ομιλία σα. Παρακαλώ, συνάδελφοι, να χειροκροτήσουμε του ομιλητέ. Και πάρα αυτά να περάσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διαταξή σα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίε και κύριοι.

Colleagues. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ καθίστε. Uh, we are going, uh, to... Να ξεκινήσουμε με το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Όπου και θα παρουσιάσουμε τη συνεργασία με τρίτες χώρες, τις αποστολές και πά. Ιδιαίτερως θα επικεντρωθούμε σε δύο παραδείγματα στις περιπτώσεις της Νορβηγίας και της Γεωργίας. Με χαρά μου λοιπόν θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω τους εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Έχουμε την κυρία Κλάρα Γκάνσλαντ, προϊστάμενη του τμήματος της ΚΕΠΑ και των σχετικών προγραμμάτων και συμφωνιών, εταιρικέ σχέσει και συμφωνίε τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ε, στη συνέχεια έχουμε την ε, πρέσβυρα Ingrid Σουλερούτ, αναπληρώτρια επικεφαλή της αποστολής τη Νορβηγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, τον κύριο Ηρακλή Κοχασβίλη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της αποστολής της Γεωργίας από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην, ε, του Υπουργείου Άμυνας, συγγνώμη. Κύριε και κύριοι, είμαστε κάπως πιεσμένοι χρονικά. Καθυστερήσαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση, συζήτηση, συγγνώμη. Αλλά το θέμα αυτό προφανώς είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και προφανώς ε, Θέλουμε να ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε. Θα θέλαμε να δώσουμε λοιπόν το λόγο στους ομιλητές. Δεν θα μακρηγορήσω. Έχετε το λόγο κυρία Γκάνσλαντ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και καλημέρα σας. Σε ευχαριστούμε για την πρόσκληση για να σας μιλήσω για, τις, ε, για την συνεργασία που έχουμε στα πλαίσια της ε, Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας με κάποιες ε, Τρίτε χώρε γειτονικέ. Καταρχήν το γενικό πλαίσιο και υπόβαθρο. Ε, με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώσαμε πέρυσι πόσο προχώρησε η συνεργασία και πώς οι εταίροι μας συνεχίζουν να στηρίζουν ενεργά την κοινή μας πολιτική ασφάλειας και άμυνας, την ΕΠΑ. Είχαμε διάλογο για την ασφάλεια και την άμυνα που διευρύνθηκε και πέρασε σε πολλά επίπεδα από διαβουλεύση υψηλού επίπεδου με τον Πέντρο Σεράνο, τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα με τους ομολόγους του, με πολλές οργανώσεις και συνεχής συζητήσεις και συνεδριάσεις σε επίπεδο υπηρεσιών. Στόχος του διαλόγου αυτού είναι σίγουρα η ανταλλαγή πληροφοριών για του τομεί δραστηριοτήτων μας και το σχεδιασμό σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, αλλά και προώθηση της ε, συνεννόησης και της αμοιβαίας κατανόησης με τους εταίρους. Ε, επίσης κάνουμε αξιολόγηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε στον τομέα της ασφάλειας και συζητούμε και προσπαθούμε να διευκολύνουμε τη συμμετοχή τρίτων χωρών στις επιχειρήσει και αποστολές μας τη ΕΠΑ. Αυτή αυτήν την άποψη, οι τρίτες χώρες ε, συνέβαλαν τα μάλα και σε επίπεδο προσωπικού αλλά και σε επίπεδο ικανοτήτων στις ε, αποστολές και επιχειρήσεις της ΕΠΑ. Για παράδειγμα, είχαμε την ομάδα ε, προστασίας από τη Γεωργία, προστασίας ε, των στρατικών δυνάμεων, EU και τώρα στο EU TMRCA. Επίσης, έχουμε τη φρεγάτα που πρόσφερε η Κορέα στην επιχείρηση Αταλάντη στήριξη επίπεδο μυστικών υπηρεσιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επιχείρησή μας Σοφία και η ιατρική υποστήριξη που παρέχει η Σερβία σε όλες τις ευρωπαϊκές αποστολές ε, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πολύ σημαντική συμβολή και της Σερβίας. Να σας υπενθυμίσω για ποιους λόγους για την πολιτική συνεργασία ε, και εταιρική σχέση της ΕΠΑ έχουμε τέτοια συνεργασία με τρίτες χώρες. Η συμμετοχή εταίρων σε επιχειρήσεις και αποστολές της ΕΠΑ και η στενή συνεργασία μεταξύ μας καταρχήν βελτιώνει την ε, διαλειτουργικότητα με τις χώρες αυτές και συμβάλλει στον επιμερισμό του άχθους της ασφάλειας. Επίσης, η συνεργασία προωθεί την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και μας, τους επιτρέπει καλύτερη ηθιγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ενδιαφέρον για τις χώρες που προσβλέπουν σε στενότερη επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης μπορεί να βοηθήσει μια τέτοια συνεργασία την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει κάποια κενά ή να αποκτήσει ειδική εμπειρογνωμοσύνη. Μάλιστα, οι εταιρική σχέση ΕΠΑ είναι και μέσο για την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασία με τρίτε χώρε, προκειμένου να αναπτύξουν και τη δική του ανθεκτικότητα και εν καιρό να βελτιώσουν και τη δική μας ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κατάσταση. Αν ε, εξετάσουμε το Μάρτιο του 2017, είχαμε 13 χώρες εταίρους που συνέβαλαν σε 9 αποστολές και επιχειρήσεις ΕΠΑ με 500 μέλη προσωπικού. Βέβαια αυτό είναι ένα απλό στιγμιότυπο γιατί δεν είναι στα πάγιο, πάγια αυτή η συμβολή. Υπάρχει μια δυναμική εξέλιξη ανάλογα με την αναλλαγή που γίνεται και ούτω καθεξής. Άλλωστε δεν είναι οι αριθμοί που μετράνε περισσότερο αλλά πώς ε, συμβάλλουν αυτές οι τρίτες χώρες στις αποστολές αυτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την EUTM-RCA, μάλιστα εκεί προσκαλέσαμε τρίτες χώρες. Στις 18 Μαΐου πέρυσι η πολιτική ασφάλειας αποφάσισε να προσκαλέσει 9 χώρες να συμμετέχουν σε αυτή την αποστολή, την EUTMRCA, μαλιστα εκει προσκαλεσαμε τριτες χωρες στις 18 μαιου περυσι η πολιτικη Ασφάλεια αποφασισε να αυτών των χωρών βρίσκεται, είναι ε, και η Γεωργία και η Νορβηγία. Και μάλιστα, όπως, είπα, όπως σας είπα, η Γεωργία συνέβαλε και με την ομάδα προστασίας ε, ε, των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα, θα ήθελα να απευθυνθώ απευθεία στον συνάδελφο από τη Γεωργία και να μιλήσω ιδιαίτερα για τη συνεργασία μας με τη Γεωργία. Θα ήθελα να εκφράσω την ε, ικανοποίησή μου για την ενίσχυση της συνεργασίας που έχουμε με τη Γεωργία σε θέματα ΕΠΑ και να εξάρω τη συμβολή της Γεωργίας της επιχειρήσης της ΕΠΑ και κυρίως στη συμμετοχή της στην ε, αποστολή εκπαίδευσης UTMRCA. Και μάλιστα έχουμε μια ε, μοίρα προστασίας ε, από τον περασμένο Μάιο, Μάρτιο. Ενθαρρύνω την Γεωργία να συνεχίσει την ε, συμμετοχή της σε τέτοιες αποστολές ε, ΕΠΑ και μάλιστα να στείλει προσωπικό και σε άλλες αποστολές και όχι μόνο σε αυτή την τελευταία τη στρατιωτική εκπαιδευτική αποστολή. Αυτό είναι αμοιβαίο υποφελές και για τις ικανότητές μας. Μάλιστα, πολλές φορές ε, ενισχύουν τις ικανότητές μας με τη συμμετοχή τρίτες χώρες, τη διαλειτουργικότητα, την απόκτηση εμπειριών, αλλά με τη συμμετοχή τρίτων χωρών ενισχύεται η νομοποίηση της ΕΠΑ, γιατί δείχνει ότι δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό όραμα, αλλά εμπλέκει και άλλους εταίρους. Σε ό,τι αφορά τον βράχη και μέσο πρόθεσμο και τις άλλες πολιτικές, θέλουμε να ενισχύσουμε, να διαβρύνουμε την συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και να δημιουργήσουμε μια ε, οικοδόμηση ικανοτήτων. Επίσης να δούμε πώς αναπτύσσουμε τις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές ε, ικανότητες μας που απαιτούνται για τέτοιες αποστολές. Φυσικά θέλουμε να ε, διατηρήσουμε τις αποστολές παρακολούθησης επιτόπου που στις 14 Δεκεμβρίου του 2018 εκπνέει η εντολή της Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της συνεργασίας μας και με τη Γεωργία. Επίσης, καλωσορίζουμε την χαιρετίζουμε την ολοκλήρωση της, ε, ε συμφωνία... της... της συμφωνίας, κάτι που θα διανοίξει νέες, ε, νέους ορίζοντες στη συνεργασία μας για την ασφάλεια. Αυτός προς τη Γεωργία. Τώρα ως προς την Ορβηγία. Φυσικά χαιρετίζουμε το ενδιαφέρον της Νορβηγίας να συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή, στις Ευρωπαϊκές Αποστολές ΕΠΑ. Πολύ σημαντικός ε, και ομοειδάτης εταίρος η Νορβηγία με κοινέ αξίες και μάλιστα εκτιμούμε ιδιαίτερως τη μακροχρόνια μας εταιρική σχέση και την υποστήριξη της ε, Νορβηγίας που συνδράμε αυτή τη στιγμή και στην ε, Συμβουλευτική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία. Είμαστε έτοιμοι και για περαιτέρω συνεργασία, προκειμένου να διερευνήσουμε και νέου τομεί συνεργασία σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, ώστε να έχουμε πιο συγκεκριμένη και απτή συνεργασία. Επίση, θα την Ορβηγία να ε, παραμείνει στις ε, αποστολές της ΕΠΑ, να διατηρήσει αμύωτη την συμβολή της και την προσκαλέσαμε και στην ε, η UTM στην εκπαιδευτική αποστολή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ε, που έχει προσκληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και καλέσαμε και την Ορβηγία. Η συμμετοχή σε τέτοιες αποστολές ε, είναι πολύ σημαντικές και δεν ε, περιορίζονται σε επίπεδο προσωπικού, αλλά έχουν και οικονομικό χαρακτήρα και πραγματικά κάνουν τη διαφορά επιτόπου σε κάποια παράλληλα σχέδια, για παράδειγμα, που ενισχύονται με τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εκπαιδευτικές αποστολές. Επίσης, ε, μας στηρίζει και στη δημιουργία ε, και στην δημιουργία ικανότητων και στην οικοδόμηση ικανότητων. Έχουμε τακτικό διάλογο σε θέματα ασφάλειας και άμυνας με την Ορβηγία επίσης, κάτι που παρέχει χρήσιμες ευκαιρίες για πιο λεπτομεριακή ανάλυση των κοινών μας αξιολογήσεων για τις προκλήσεις της ασφάλειας και τις δυνατότητες συνεργασίας. Επίσης, μη ε, ευρωπαϊκή χώρα, χώρα ΝΑΤΟ, ανήκει η Νορβηγία σε μια ειδική ομάδα ε, με την οποία συμμετέχει με ειδική σύνθεση η, Επιτροπή Ασφάλειας και επίσης ε, η Στρατιωτική Επιτροπή συνεδριάζει με αυτή την ειδική σύνθεση συν 7 και υπάρχει και μια άλλη σύνθεση συν 9. Πάντως και με την Επιτροπή την πολιτική ασφάλεια ε, ε, συνεργαζόμαστε με την Νορβηγία και τους συμμάχους μας του ΝΑΤΟ. Και σε τέτοιου είδου συνεδριάσεις, είχαμε μια τέτοια ε, συνεδρίαση ΣΥΝ 7 το 2016, κάτι που μας έδωσε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για θέματα ασφάλειας και άμυνας όπως οι κρίσεις στη Λιβύη και τη Συρία. Λυπάμαι που μακρηγόρησα, αλλά ήθελα να καλύψω πολλά θέματα, γιατί πραγματικά εκτιμούμε ιδιαίτερο στη συνεργασία με τις χώρες αυτές. Ευχαριστούμε. Να δώσω τώρα το λόγο στον, στην πρέσβη Σούλερουντ. Αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, σας ευχαριστώ πολύ για την αδότητα αυτή του διαλόγου σήμερα για τη συζήτηση μαζί σας. Είναι τιμή και χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα, μια γενικότερη νορβηγική προοπτική. Προτού πάω στις επιχειρήσεις ΚΕΠΑ. Θα ήταν χρήσιμο πιστεύω. η Νορβηγία έχει μια ευρύτατη συνεργασία επί θεμάτων αμυντικής πολιτικής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια συνεργασία που τη θεωρούμε πολύτιμη και θέλουμε να την ενισχύσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι λοιπόν που αυτές οι κοινέ επιχειρήσεις ΚΕΠΑ ε, θα μπορούσαν να είναι εξαιρετικά σημαντικές για τις πρώιμες φάσεις ε, του σχεδιασμού αντιμετωπίζουμε όλο και πιο σημαντικές και άμεσες προκλήσεις. Ζούμε σε ταραχώδεις καιρούς και νομίζω ότι ο βασικός δεσμός, ο ατλαντικός δεσμός θα παραμείνει βασικός πυλώνας αμυντικής πολιτικής. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερη ευρωπαϊκή συνεργασία και όχι λιγότερη για να τα καταφέρουμε αυτά. Εμείς είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής μέσω του ΑΣΑ μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχουμε άμεσες ε, σχέσεις ε, μέσω και της ε, περιοχής Σέγγεν, της σχέσης Σέγγεν, της κοινή δομής της ΚΕΠΑ, στα θέματα Τζάι, στα θέματα τα εσωτερικά και τα αμυντικά. Είμαστε ένας εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα αυτά τα επίπεδα. Εχθές είχαμε τον Υπουργό Αμήνης που επισκέφθηκε την ΙΕΔ και σήμερα ο Υπουργός Μπρέντα ε, συζητά με την κυρία Μογκερίνη για μια, σε μια επιτροπή ad hoc για θέματα που αφορούν στην Παλαιστίνη. Είχαμε συναντήσει με τον κύριο Τους και τον κύριο Γιούνκερ, δηλαδή ο διάλογος που διεξάγεται μεταξύ Νορβηγίας και Αρακής Ένωσης είναι απολύτως ε, ε, τακτικός και συστηματικός και σε όλα τα επίπεδα. Στα επόμενα 7 χρόνια θα συνεισφέρουμε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου μέσω του, ε, των κοινών προγραμμάτων στήριξης στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και θα ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ Νορβηγίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης επί θεμάτων ασφάλειας όπως λέει και η Λευκή Βίβλος οι, οι στοχεύσεις ε, ε, ευημερίας και ασφάλειας είναι κοινή έχουμε μεγάλες θαλάσσιες περιοχές, ενεργειακούς πόρους, ε, θαλά... Ε, ε, αλλιευτικά αποθέματα, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε επίσης χερσαία και θαλάσσια σύνορα με την Ρωσία, που είναι ένας μεγάλος γείτονας και απρόβλεπτος συχνά. Όλα αυτά διαμορφώνουν λοιπόν την πολιτική μας, την αμυντική και ασφαλείας. Είχαμε λοιπόν ένα πρόσφατα εγκρίνει ένα αμυντικό σχέδιο για το 2017 με μακροπρόθεσμο στόχο να προσθέσουμε περί τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ στον προπολογισμό των αμυντικών, δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων για τα επόμενα 20 έτη. Αυτό είναι ένα ασφαλές μήνυμα ότι η Νορβηγία λαμβάνει τις δεσμεύσεις της αμυντικές πάρα πολύ σοβαρά. Ο ακρογωνίας λήθος της ε, αμυντικής μας πολιτικής είναι το ΝΑΤΟ και όπως είναι και για τις περισσότερες ορακίες χώρες. Η εστίασή μας στην διατλαντική σχέση κατευθύνει την πολιτική μας εδώ και δεκαετίες και θα εξακολουθήσει να το κάνει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Και μπορούμε να βοηθήσουμε τις εταίρες μας σε πάρα πολλά σχετιζόμενα αμυντικά θέματα. Χαιρετίζουμε λοιπόν κάθε πρόταση ενίσχυσης της συνεργασίας και της διατηρητικής αυτής σχέσης και θεωρούμε ότι αυτή θα είναι αμοιβαία υποφελής για τα θέματα ασφαλείας και άμυνας. Έχουμε κοινέ αξίες, αλλά έχουμε διαφορετικά μέσα στη διάθεσή μας, τα οποία όμως είναι πολύ συχνά αλληλοσυμπληρωματικά. Μπορούμε να συζητήσουμε περαιτέρω νορβηγική εισφορά σε θέματα, σε περιοχές όπου θα συμφωνήσουμε από κοινού, όπως οι βρετικές απειλές, οι θαλάσσιες απειλές, η άμυνα στον κυβερνοχώρο και βεβαίως η αντιμετώπιση της τρομοκρατία. Έχουμε λοιπόν ένα περιβάλλον όλο και πιο περίπλοκο με απειλές ε, και κίνδυνο διεθνώ. Ε, έχουμε ε, πολύ συχνά διάφορες κρίσεις και πολεμικές ζώνες στην ευρύτερη περιφέρεια της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμπεραίνουμε και στην Νορβηγία όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η προάσπιση της ασφάλειάς μας πρέπει να πηγαίνει πολύ πέρα από τα σύνορα τα ευρωπαϊκά. Πρέπει να εξασφαλίσουμε καλύτερη διάδραση και συντονισμό μεταξύ των μέσων ε, πολιτικής κέπα που είναι διαθέσιμα σε εμάς. Την περασμένη εβδομάδα η νορβηγική ε, κυβέρνηση παρουσίασε τη νέα λευκή της βίβλο για την νορβηγική ε, εξωτερική πολιτική με βασικό πόρισμα ότι πρέπει να εντατικοποιηθεί η συνεργασία της Νορβηγίας με τις ευρωπαϊκές χώρες και τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας ε, στον, στην ε, περιοχή του Νότου και της Ανατολής της Ευρώπης ενισχύοντας και τη Διατλαντική Συμμαχία. Θα υλοποιήσουμε τη στρατηγική για να ενισχύσουμε ευάλωτα κράτη ε, στην Βόρεια Αφρική και στο Σαχέλ θα ενισχύσουμε την παρουσία μας στην περιοχή και θα αυξήσουμε τη στήριξή μας προς συγκεκριμένες χώρες ε, στο Μαλί, την, ε, την Ισία, στο Μαρόκο. Θέλουμε να δούμε πιο στενή συνεργασία αμυντική με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη φάση του σχεδιασμού και στη φάση της υλοποίησης. Κοινών αποστολών δηλαδή και ΕΠΑ. Η Νορβηγία συνεισφέρει ως εταίρος σε διάφορες τέτοιες αποστολές πολιτικής και στρατιωτικής φύσεως από το 2002. Το 2004 συνυπεγράφει ένα εταιρικό πλαίσιο που προβλέπει τις διαδικασίες ε, της συμμετοχής της Νορβηγίας σε τέτοιες κοινέ αποστολές. Αυτό το κάνουμε κατά περίπτωση και η συμφωνία αυτή πλαίσιο ε, συνεισφέρει στην ομαλή υλοποίηση των επιμέρους ε, ρητρών. Όλα αυτά βεβαίω σημαίνουν πολύ σημαντική ευθύνη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις συνεισέρουσες χώρες. Ιδιαίτερα στην περίπτωση τρίτων χωρών χρειάζεται έγκαιρος συντονισμός, χρειαζόμαστε πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες και για στρατηγικές αναλύσεις αλλά και για πρακτικής φύσεως αναλύσεις εγκαίρως ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε τις ε, σωστές αποφάσεις συμμετοχής ή όχι. Η έγκυρη αυτή ενημέρωση είναι επίσης απαραίτητη και κοινοβουλευτικά, κάτι το οποίο είμαι βέβαιο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατανοεί πλήρως. Θα θέλαμε λοιπόν μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα στις πρώιμες φάσεις σχεδιασμού. Η Νορβηγία ως κράτος μη μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συμμετέχει στην διαδικασία λήψης απόφασης και επομένως πρέπει να έχει απόλυτη ενημέρωση. Ένα ένας τρόπος να επιλύσουμε το ζήτημα αυτό θα ήταν να διευρύνουμε την Επιτροπή Εισφορέων ώστε να συμμετέχει και στη φάση του σχεδιασμού και υλοποίησης. Πρέπει να υπάρχουν και άλλοι τρόποι ώστε τρίτες χώρες να συμμετέχουν σε αποστολές παρά μόνο και μόνο μέσω της εισφοράς προσωπικού. Υπάρχει ηλική βοήθεια, υπάρχει οικονομική βοήθεια και άλλα είδη βοήθειας. Αυτό θα δώσει έναν ευέλικτο τρόπο σε χώρες που θέλουν να συνεισφέρουν και θα, θα συμβάλλει σε μια καλύτερη κατανομή του όλου φόρτου. Έχουμε συνεισφέρει σε αποστολές όπως το Κόσοβο, στην Ινδονησία, στον ε, κόλπο της Αντέν, για να αναφέρω μόνο μερικές, και γνωρίζουμε ότι έχει εκτιμηθεί η συνεισφορά μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, όπως και τις χώρες που φιλοξενούν τις αποστολές. Και όλη αυτή η εμπειρία είναι πολύτιμη που μας φέρνουν δηλαδή οι συμμετέχοντες Νορβηγοί εμπειρογνώμονες πίσω στη χώρα. Η συμμετοχή μας σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι η πιο εμφανής συμμετοχή μας στον, στα θέματα ΚΕΠΑ. Η Νορβηγία θα εξακολουθεί να διεκδικεί έναν ενεργητικότατο ρόλο στα θέματα αυτά. Και είμαστε ανοιχτοί και σε νέα πεδία συνεργασίας επιθεμάτων ευρύτερα συνδεδεμένων με την ΚΕΠΑ. Όπως ανέφερε και η ΕΔ, το PFC συν 7 και συν 9 θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο ανταλλαγής. Υπάρχουν και άλλα επίπεδα, όπως οι στρατιωτικές επιτροπές, και χαιρετίζουμε και την διαβούλευση και με τρίτες χώρες ή στο πλαίσιο των στρατιωτικών αυτών αναλύσεων. όλες αυτές οι αναλύσεις ε, και εκθέσεις είναι πολύ σημαντικές για εμάς και θα θέλαμε να συμβαίνουν πιο τακτικά και πιο συχνά. Τελικώ ήθελα να πω ότι χαιρετίζουμε τι προσπάθειε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτυχθεί μια στρατηγική, στρατηγική προσέγγιση μεταξύ τη Ένωση και των χωρών εταίρων στα θέματα εξωτερική πολιτική και πολιτική αμήνη Γνωρίζω ότι πολλά από αυτά τα θέματα που ανέφερα συζητώνται ήδη στα πλαίσια αυτής της ε, προσπάθειας και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Υπό τη δική μας οπτική γωνία αυτό ευθυγραμμίζεται απολύτω με την ε, έμφαση στην συνεργασία με τρίτες χώρες στη Λευκή Βίβλο. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας και τη διαβούλευσή μας με τους Ευρωπαϊκούς ώστε να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε στο τεράστιο δυναμικό που υπάρχει στην κοινή μας εταιρική σχέση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρα, για την ε, συνεκτικότατη αυτή ενημέρωση σε ό,τι αφορά το νορβηγικό σύστημα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση και σα ακούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ηρακλή Κορασφίλη από τη Γεωργία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα και σε όλους. Καλημέρα αγαπητοί βουλευτές, μέλη της Επιτροπής. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω για την εμπειρία μου αυτή στην συμμετοχή στην αποστολή στην ΚΕΠΑ. Θα ήθελα να παρουσιάσω το υπόβαθρο της αποστολής αυτής και να δώσω κάποια θετικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην αποστολή αυτή και κάποια πορίσματα τα οποία έχουμε ε, να εξαγαγούμε. Θα γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωποίηση είναι μία ένωση πολιτικής συνενέσεις και ε, υποστήριξης. Η Γεωργία λοιπόν είναι δεσμευμένη στην ατζέντα συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γεωργίας και έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή για την τόνωση της ευρωπαϊκής προοπτικής. Μεταξύ των κυρίων προτεραιοτήτων μας συγκαταλέγεται λοιπόν και η εμβάθυνση της συνεργασίας το τομέα της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, ιδιαίτερα και αυτή η συμμετοχή σε απόστολες και πά. Αυτό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της, ευρωπαϊκής γεωργιανής ατζέντα. και αυτό για διάφορους λόγους. Είμαστε πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε αυτές τις αποσχόλες για διάφορους λόγους. Καταρχάς, αισθανόμαστε ότι είμαστε μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας και θέλουμε να συμμετέχουμε στην κοινή οικοδομήση της ε, ασφάλειας. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι ακεραιοί και ε, ε, ανεξάρτητοι και ελεύθερη η Ευρώπη σε ό,τι αφορά τώρα την αλληλοσύνδεση που υπάρχει και την αλληλοεξάρτηση σήμερα και από γεωγραφικής άποψης. Άρα πιστεύουμε ότι όλα αυτά κινούνται πέρα από τα σύνορά μας και ο τρίτος λόγος ήμασταν ατυχείς σε ό,τι αφορά την επίθεση των βορειών γειτόνων μας. Αυτό λοιπόν οδήγησε σε διάφορες καταστάσεις στη Γεωργία και θα ήθελα να... Και τώρα πλέον θέλουμε να πετύχουμε τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή αυτή. Είμαστε ευγνώμονε λοιπόν για τη συμμετοχή και τη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε και εμεί να ενισχύσουμε με τη σειρά μα την ασφάλεια και στην περιοχή μας αλλά και πέρα από την περιοχή μας. Η Γεωργία έχει αποδείξει επανελειμμένα ότι δεν αποτελεί μόνο καταναλωτή της ασφάλειας, αν θέλετε, αλλά και πάροχο της ασφάλειας, ε, σύμφωνα και με τη Διεθνή Σύμβαση του Ελσίνκη. Και τέλος, τελευταίος λόγος, αλλά και πολύ σημαντικός, είναι ότι η συμμετοχή σε τις αποστελές ε, ΚΕΠΑ είναι μια πάρα πολύ σημαντική εμπειρία από πλευράς ε, ναι, συγγνώμη λέει η πρόεδρο που σα διακόπτω. Αν θα μπορούσατε να μιλάτε λίγο πιο αργά, γιατί ενδεχομένω να έχουν προβλήματα διερμηνή. Και ο τελευταίο λοιπόν λόγο τον οποίο και αναφερόμουν, ε, επιτρέπετε μου να επαναλάβω, είναι ότι η εμπειρία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Συλλέγουμε σημαντικέ εμπειρίε από τη συμμετοχή σε τέτοιε αποστολέ και πά. ενισχύει αυτό τις στρατιωτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων της Γεωργίας και προωθεί και την διαλειτουργικότητα των στρατιωτικών δυνάμεων μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Οι ένοπλες δυνάμεις της Γεωργίας έχουν σημαντική εμπειρία σε συμμετοχή σε διάφορες αποστολές για την διατήρηση και την επιτεύξη της ειρήνης από αποστολές από το 1999 και μετά. Ο Πέρσικος κόλπος Βαλκάνια, Αφγανιστάν το 2013 υπογράψαμε και μια συμφωνία πλαίσιο συμμετοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελεί και τη νομική βάση για την δέσμευσή μας και τη συμμετοχή μας σε τέτοιες αποστολές και πά. Από το 2014 και εφ' ε, για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2014 αναπτύξαμε τα στρατεύματά μας στο ε, U4RCA. Θα ήθελα λοιπόν να σας υποδείξω στο σημείο αυτό να επιστήσω την προσοχή σας στο εξή ότι έχουμε ανα... αναπτύξει τέτοια τέτοιες. Έχουμε χρησιμοποιήσει 156 τέτοιες εταιρείε για την ανάπτυξη τέτοιου στρατευμάτων. Και η συμμετοχή αυτή ε, δεν περιορίζεται στην ολοκλήρωση των αποστολών. Συνεχίζεται και μετά. με δύο μοίρε και στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Συνεχίζουμε την συμμετοχή μας με πέντε ομάδες άμεσης ανταπόκρισης και πλέον έχουμε μία δημιουργία και δεσμευόμαστε να παραμείνουμε στην αποστολή μέχρι το τέλος της, ε, του UNTRCA, της στρατηγικής αυτής επιχείρησης. Ε. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή από πλευρά της Γεωργίας. Να σας ευχαριστήσω όλους και να ευχαριστήσω και την κυρία Γκάντσλαντ για τα βιανικά της λόγια για την ε, συμβολή μας. Τώρα, να βράσω στο επόμενο θέμα. Αναφέρθηκα στη συμμετοχή λοιπόν σε αποστολές και στο UTN Mali στη θεσμική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι ε, συμμετέχουμε μέχρι το 2018 το Μάιο προβλέπεται η αποστολή αυτή και τέλος με περηφάνεια να σας αναφέρω ότι καταφέραμε να συμμετέχουμε και στην αποστολή πολιτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στην Ουκρανία από το 2014 με εμπειρογνώμονες για πλέον του ενός έτους. Και νομίζω ότι πολλά μαθήματα εξάγαγαμε από τη συμμετοχή αυτή της Αποστολής. Να σας αναφέρω ότι αντιμετωπίσαμε και κάποιες προκλήσεις σε ό,τι αφορά τις αποστολές και πα, προφανώ. Αλλά χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την αμέριστη υποστήριξη από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο σε ό,τι αφορά τι αποστολές αυτές επιτόπου. Και θα ήθελα επίσης να αναφέρω για ένα καταπίστευμα για την ΚΕΠΑ, το οποίο διαχειρίζονται οι λιθιονικέ αρχές. Αντιμετωπίζαμε προβλήματα, θεωρούμε τα προβλήματα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς και έτσι συνεχίζεται η συμμετοχή μας σε ό,τι αφορά τη φύση των αποστολών και πά. Το βασικό πρόβλημα, ξέρετε, είναι η χρονική περιορισμοί. Οι χρονικοί περιορισμοί για την ε, κατάρτστρωση και την ανάπτυξη των σχεδίων. Ε. Και αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο για τρίτες χώρες, ξέρετε γιατί σε πρώτη φάση θα πρέπει να ληφθεί και η πολιτική απόφαση κατά πόσο υπάρχει η πολιτική βούληση για τη συμμετοχή στην αποστολή. Μετά υπάρχει και όλη η διαδικασία από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να αξιολογηθεί η πρόσφορά μα, να δοθεί α, συνένεση για την συμμετοχή μα και μετά έχουμε τι τεχνικέ, το τεχνικό σκέλο και το νομικό σκέλο. Και όλα αυτά φυσικά είναι χρονοβόρα, προκαλούν καθυστέρηση τη ανάπτυξη ε, των δυνάμεών μας και ένα σημαντικό πρόβλημα για τα γεωργιανά στρατεύματα είναι η στρατηγική υποστήριξη και η υποστήριξη επιμελητίας επιτόπου, γιατί η δυνατότητα πρόβλεψη των δυνάμεων που θα χρειαστούν είναι πολύ περιορισμένη. Έτσι γίνονται λοιπόν διμερείς διαβουλεύσει, υπάρχει υποστήριξη από το CMPD UMS. Όλα αυτά λοιπόν ως σκοπό έχουν να εντοπίσουν ενδεχόμενους παροχούς βοήθειας και αυτό προφανώς με τη σειρά του καθυστερεί και την ανάπτυξη των δυνάμεων μας. Υπήρξε λοιπόν ε, και κάποιες δυσκολίες οι οποίες παρεμπόδισαν την ε, ομαλή εκτέλεση της αποστολής επιτόπου αλλά θα επαναλάβω στο σημείο αυτό και θα υπογραμμίσω εκ νέου ότι καταφέραμε να ε, αντιμετωπίσουμε με επαγγελματικό τρόπο τις δυσκολίες και με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού προσωπικού, της προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τέλος, να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει διαρκής υποστήριξη του κοινού για τις ευρωπαϊκές αυτές αποστολές και προς την κατεύθυνση αυτή. Κάνουμε δημόσιες ε, ενημερωτικές εκστρατείες για ενημέρωση της, του κοινού ε, για τις αποστολές αυτές. Φιλάνδια, μέσα ενημέρωση, κοινωνικά μέσα και το πρόβλημα είναι σε ό,τι αφορά την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας ότι τα σημαντικά επιτεύγματα η βίζα ε, εκείνη η ατζέντα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γεωργίας όλα αυτά υποστηρίζουν και προφανώς δίνουν έναυσμα για να συνεχίσει το κοινό να υποστηρίζει με τη συμμετοχή μας σε τέτοιες αποστολές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε λέει και η Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χασβίλη για την παρουσίαση αυτή και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής για να γίνει η συζήτηση. Ο κύριος Γκάλερ θα θέλει να πάρει το λόγο. Ναι, ενδιαφέρον γιατί για δεύτερη φορά πρέπει να ξαναζητήσω συγγνώμη που έχασα τις ε, αρχικές παρεμβάσεις. Αλλά δυστυχώς συμπίπτουν πολλές συνεδριάσεις και τρέχουμε αριστερά και δεξιά. Ήμουνα στην στο τελευταίο τμήμα τη εβδομάδα τη Τινησίας ε, που είχαμε αυτή τη βδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί η Τινησία είναι και στη νότια γειτονία και είναι πολύ κοντά σε περιοχές κρίσεων και ίσως επίσης ε, θα μπορούσε να είναι υποψήφια για συμμετοχή και συνεργασία σε αποστολές και πά. Έτσι να προωθήσω και αυτή την ε, χώρα. Χαίρομαι πάντως ε, για την παρουσία εκπροσώπων της Νορβηγία και της Γεωργίας. Ε, καταρχήν η, Γεωργία, η Νορβηγία είναι πλήρες μέλος ΝΑΤΟ του Σέγγεν, του ΕΟΧ και είναι από πολλές απόψεις πολύ κοντά μα η Νορβηγία και πρόσκειται ε, σε μεγάλο βαθμό στις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάνει ένα επιπλέον βήμα συμμετέχοντας σε αποστολές και επιχειρήσεις και πά. Σε ό,τι αφορά τη γεωργία, είχα πάει δύο φορές στη Γεωργία. Μία ήταν σε αποστολή μάλιστα της υποεπιτροπής ε, μας ΣΕΝΤΕ και σε μία αποστολή παρατήρηση εκλογών ε, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ε, παρατηρήσαμε το φαινόμενο της συνοριοποίησης, όπως λέμε, των κατεχόμενων εκεί. Και χαίρομαι που η Γεωργία συμμετέχει ενεργά και συμβάλλει τόσο σημαντικά στις αποστολές και πά. Και είναι ένας καλός προάγγελος ε, των περαιτέρω βημάτων ε, για πιο στενή συνεργασία και σύνδεση. Ξέρετε πως λειτουργούν αυτά τα πράγματα και πραγματικά είναι χρήσιμη η συνεργασία μας ε, γιατί εξακολουθεί να διατρανώνει τις αμοιβέ ε, δεσμεύσεις για τέτοια στενή συνεργασία. Θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Γεωργίας αν η χώρα σας είναι ικανοποιημένη από το βαθμό συνεργασίας, δηλαδή ε, πώς βλέπετε την κατάσταση επιτόπου, σας βοηθά αυτή η συμμετοχή, μήπως σας ε, επιβαρύνει υπερβολικά ως προς τις οικονομικές πτυχές. Τι γίνεται, γιατί δεν ξέρω αν προβλέπονται ειδικέ διατάξεις πέραν του μηχανισμού Αθήνα για τη χρηματοδότηση αυτών των ε, αποστολών. Ε, ισχύει το ίδιο και για σας υπάρχουν άλλες ειδικέ διατάξεις για τη Γεωργία. Πώς έχει ειδικά η κατάσταση για την Νορβηγία. <laughs> για την Νορβηγία δεν έχω καμία αμφιβολία ότι έχει τη δυνατότητα την οικονομική να συμμετέχει σε τέτοιες αποστολές και δεν χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση. Σας ευχαριστώ. Κύριο Στέτινα. Βάλτε παρακαλώ τα ακουστικά σας γιατί θα μιλήσω τσεχικά. Ε, ε, Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Καχασβίλη και ο λόγος που τη θέτω είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα μεταβώ στην Τυφλίδα ως μέλος της αντιπροσωπείας ε, του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συζητήσουμε με την Γεωργία ζητήματα ασφάλειας. Είπατε ότι αποσπάσματα με γεωργιανούς στρατιώτες, οι γεωργιανές δυνάμεις συμμετέχουν σε αποστολές και ΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω όμως και έναν άλλο τομέα συνεργασίας. Ξέρω ότι στην Ουκρανία υπάρχει ένα ε, τάγμα εθελοντών από τη Γεωργία στην ε, κοιλάδα Ντονέτσκ Ξέρω ότι στις, ε, στα τάγματα αυτά συμμετέχουν και γεωργιανοί στρατιώτες όπως ε, και ευρωπαίοι στρατιώτες. Δεν είναι όμως ε, επίσημοι εκπρόσωποι των χωρών, είναι θελοντές που πηγαίνουν και ο θελός και συμμετέχουν σε αυτό το τάγμα βοηθώντας την Ουκρανία να αντιταχθεί σε αυτή την ρωσική επίθεση στον Ντονέτσκ στην κοιλάδα Ντομπάς. Η Γεωργία έχει και επίσημα λάβει μέρος σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Δηλαδή έχει συμπαραταχθεί και επισήμως ε, στο πλευρό της Ουκρανίας ε, έναντι αυτής της ρωσικής επίθεσης και Υπάρχει κάποια στρατιωτική βοήθεια που προσφέρει η Γεωργία στην Ουκρανία. Γιατί Ξέρω ότι παρά το εμπάργο γίνεται εξαγωγή όπλων προς την Ουκρανία πέραν των εθελοντών στρατιωτών που συμμετέχουν σε αυτό το τάγμα. Υπάρχει άλλου είδους επίσημη συνδρομή της Γεωργίας προς την Ουκρανία. Ευχαριστώ κύριο Σκούσο. Ευχαριστώ. Εγώ θα μιλήσω ισπανικά. Θα ήθελα να ρωτήσω την ε, προϊσταμένη του τμήματος την κυρία Κάνσλαντ ε, γνωρίζουμε τα ζητήματα της ε, Νορβηγίας και της ε, Γεωργίας. Υπάρχει πρόθεση να συμπεριληφθούν και άλλες χώρες ε, σε τέτοιου είδους αποστολές και επιχειρήσεις και ΕΠΑ. Και δεν είναι παράδοξο που συμμετέχουν τρίτες χώρες όπως η Γεωργία, ενώ έχουμε από το 2008 μία αποστολή μας στη Γεωργία ε, δεν είναι από τη, παράδοξο που από τη μία ε, η χώρα είναι αποδέκτης ευρωπαϊκής αποστολής και από την άλλη η χώρα αυτή συμμετέχει σε ευρωπαϊκές αποστολές σε τρίτες χώρες. Ευχαριστώ, δεν ξέρω αν ο κύριος Ντρογεύσκη θα ήθελε το λόγο. Μάλιστα, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα θα ήθελα να εκφράσω την ε, ικανοποίησή μου για αυτήν την ευρυθή και εκτεταμένη συνεργασία με χώρες εταίρους όπως η Νορβηγία και η Γεωργία. Για μένα η Γεωργία είναι πολύ σημαντική χώρα και ο τομέας αυτός της συνεργασίας θα διδραματίσει κέριο ρόλο για την σταθεροποίηση της πολιτικής και στρατιωτικής κατάστασης σε μια τόσο δύσκολη γεωγραφική περιοχή. Σας ευχαριστώ θερμά λοιπόν που περιλάβατε αυτό το θέμα σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Σε ό,τι αφορά την Νορβηγία, ως Υπουργό Πολιτισμού είχα πολύ θετική εμπειρία από τη συμμετοχή της ε, Νορβηγίας στη διαφύλαξη της ε, πολιτιστικής κληρονομιάς στην Πολωνία. Και αυτό ήταν ε, πολύ σημαντική και ποιοτική συνεισφορά εκ μέρους της Νορβηγίας και χαίρομαι που σήμερα η Νορβηγία συμμετέχει και σε ζητήματα και επιχειρήσεις ασφάλειας και άμυνας. Θεωρώ ότι δεν έχουμε αξιοποιήσει το έπακρο αυτή αυτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Πιστεύω ότι μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία και να προβάλλουμε τέτοιου είδους δυνατότητες διευρύνοντάς τις και ενισχύοντάς τις ταυτόχρονα. Σε ό,τι αφορά τη Γεωργία, έχω μια ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της Γεωργίας, τον κύριο Κοχασβίλη. Είναι γνωστό ότι η Γεωργία έχει δύο πολύ σημαντικού ε, αποστρεπτική άποψη γείτονε: ε, βορείως ε, τη Ρωσία και νοτίως την Τουρκία. Σήμερα πώς αντιμετωπίζετε στη Γεωργία την κατάσταση στην Τουρκία, από άποψη ασφάλειας, πώς βλέπετε τις νέες εξέλιξεις στην Τουρκία. Και τέτοιου είδους ε, ε, διάβλους επικοινωνίας δεν θεωρείτε ότι θα ε, έχουν κέρια σημασία και για τη συνεργασία στο ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να αναφέρω ότι χθες είχαμε την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων με τον Γιώργο Στόλτεμπεργκ, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. που ήρθε και μας μίλησε σε αυτή την κοινή σε ΑΦΕΤ Σέντε. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ μας παρουσίασε και τους νέους τρόπους συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Βαρσοβίας. Εσείς κύριε Πρέσβη, θα μπορούσατε να μας πείτε, ε, κυρία Πρέσβη μάλλον, τι συνεργασία περιμένει περαιτέρω η Νορβηγία πέραν των αποστολών ε, ΚΕΠΑ, όπου εκτιμούμε ιδιαίτερα στη συμμετοχή της Νορβηγίας σε επιχειρήσεις και αποστολές ΚΕΠΑ, αλλά ε, στα πλαίσια του υβριδικού πολέμου που γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα βλέπατε συνεργασία με την, της Νορβηγίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ε, και με την Ουκρανία είχαμε επάφη με προσώπους για την ε, διεξαγωγή των αποστολών, των στρατικών αποστολών και είχαμε συνεργασία με τη Γεωργία στην ε, αποστολή ΣΕΝΤΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία το 2015. Εκεί είχαμε ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους της Γεωργίας στην αποστολή αυτή, αλλά και στο παρελθόν επισκεφτήκαμε και τη στρατιωτική μας επιχείρηση στο Μαλί εκτιμήσαμε ιδιαίτερο στην συμβολή της Γεωργίας στην ε, αποστολή και πά που ήταν αναπτυγμένη στο Μάλι. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους καλεσμένους μας και να τους ξαναδώσω το λόγο για να σχολιάσουν τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Θα μπορούσαμε ίσως να ξεκινήσουμε από την κυρία Γκάρσλαντ και μετά θα ακούσουμε την Περέζ Βισούλαρουτ και στο τέλος τον κύριο Κοχασβίλη. Με την ίδια σειρά δηλαδή που μίλησαν και προηγουμένως οι καλεσμένοι. Ε, thank you, Madam. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, μπερδέψαμε τα ακουστικά μας. Σχετικά με την ερώτησή σας κατά πόσον θα προσκαλέσουμε και άλλες χώρες, ήθελα να θυμίσω ότι ήδη έχουμε 18 από αυτές τις συμφωνίες ε, πλαίσιο εγκατεστημένες αναφέρθηκαν και από τους δύο ομιλητές εδώ στο βήμα οι οποίες είναι ενδείξεις μιας επιθυμίας εκατέρωθεν των συνυπογραφόντων δηλαδή δυνατοτήτων ευρύτερης νεασίας Διευκόλυνση δηλαδή πρόσκληση σε συγκεκριμένε αποστολέ. Αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι το να έχει κανεί συμφωνία πλαίσιο δεν σημαίνει ότι είναι αυτόματα όλα τα υπόλοιπα. Κάθε φορά λαμβάνεται απόφαση ad hoc από την Επιτροπή Ασφαλείας, από το κράτος μέλος, για το κατά πόσον θα προσκληθεί η συγκεκριμένη τρίτη χώρα, για το κατά πόσον θα υπάρξει ή όχι συνεργασία Μερικές από τις αποστολές μας είναι μόνο για κρατημέλη και ακόμα και αν έχει υπάρξει προσφορά πρέπει να γίνει δεκτή κατόπιν συστάσεως των επικεφαλής, των διοικητών. Πρόκειται λοιπόν για μια ολόκληρη διαδικασία, αλλά βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα. Έρχομαι τώρα στο συγκεκριμένο ερώτημα σχετικά με την, με την αποστολή, με την φιλοξενία της αποστολής της Εβραϊκής στη Γεωργία και την συμμετοχή της σε αποστολές ΚΕΠΑ. Ε, δεν υπάρχει κάποιο, κάποια αντίφαση εδώ, κάποιο παράδοξο. Δεν είναι μόνο καταναλωτής αλλά και πάροχος ασφαλείας η Γεωργία όπως είπε και ο συνομιλητής. Εμείς εκτιμούμε την εμπειρία που έχει η Γεωργία από την συμμετοχή σε άλλες ειρηνευτικές αποστολές όπως και την συγκεκριμένη μονάδα που παρήχε. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αντίφαση σε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, η πρέσβης, να ξεκινήσω, Πρόεδρε, ευχαριστώντας τα μέλη και να πω ότι εκτιμούμε τη συνεργασία σας, τη συνεργασία με όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Για το συγκεκριμένο ερώτημα που έγινε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ε, και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, δεν μπορώ να είμαι πιο συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή, αλλά με χαρά θα επανέλθουμε σε λεπτομέρειες εμπίπτουν οι περιοχές αυτές στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λευκή βίβλος ε, που υπευλήθη στο Κοινοβούλιο της Νορβηγίας διευκρινίζει το έδαφος, το πεδίο αυτής της κοινή ε, συνεργασίας και όταν θα έχει εγκριθεί θα επανέλθουμε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Καχασβίλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και να ευχαριστήσω για τις ε, πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όλες. Καθότι προέρχομαι από τα αμυντικά θέματα ίσως θα είχα μια επιφύλαξη να πάω σε βαθύτερα πολιτικά ζητήματα. Σχετικά με την ε, χρηματική πτυχή της συμμετοχής μας σε αποστολές σε ΚΕΠΑ, θα ήθελα να αναφέρω ότι όλος ο μηχανισμός λειτουργεί αρκετά καλά ο μηχανισμός Αθένα δηλαδή και συνολικά το σύστημα συνεισφοράς μας, αλλά και το καταπίστευμα που διαχειρίζεται από τη λιθουανική πλευρά και έχει αναλάβει την οικονομική ευθύνη εις ό,τι αφορά σε δραστηριότητες υπό την ΚΕΠΑ. Όπως ελέγχθη, υπογραμμίζω και εγώ ότι σε καιρούς ε, λιτότητος και δημοσιονομική πειθαρχία αυτό περιορίζει τις ε, εισφορέ μας αλλά σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή και προχωρώ στα σχόλια του κυρίου Στετίνιους που θα μας επισκεφθείτε στην Τυφλίδα πολύ σύντομα. Με χαρά θα σας υποδεχθούμε και πάντοτε καλωσορίζουμε όλους τους φίλους ε, στη Γεωργία και όχι μόνο τους φίλους λέει ο μιλητής. Σχετικά με τη σχέση μας με την Ουκρανία, είχαμε φιλικές σχέσεις ε, επιμακρών. Δεν υπάρχει επίσημη στρατιωτική βοήθεια, ούτε ανεπίσημη, προς την Ουκρανία. για την αντιμετώπιση δηλαδή της ρωσικής παρέμβασης. Έχουμε μία συνεργασία που συμπεριλαμβάνει προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και περιορίζεται σε αυτά. Να αναφέρω ότι είχαμε συμμετάσχει ε, στην επιχείρηση ΚΕΠΑ και ο επιτετραμένος του Υπουργείου Αμήνης ε, είχε συμμετάσχει στην επίσκεψη στην Ουκρανία. Αυτό ήταν μια πολύ θετική εμπειρία. Πέραν αυτού δεν μπορώ να σας υποβάλω κάποιο άλλο σχόλιο για μυστική ή ανεπίσημη ή άλλου είδους συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις ε, γεωργιανών ή στην Ουκρανία. αλλά σας ευχαριστώ και για αυτή την παρατήρηση και προχωρώ στο θέμα το σχετικό με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι στρατηγικός μας εταίρος και από τους μεγαλύτερους, σημαντικότερους εισφορείς μας στην αμυντική μας δηλαδή ικανότητα συνολικά συνεργαζόμαστε ενεργώς από την ανεξαρτησία μας από δεκαετία του 90 μας έχουν υποστηρίξει σε διάφορα επίπεδα και πολύ συγκεκριμένα στο επίπεδο της αμήνης και των ενόπλων δυνάμεων. Πρόκειται για μια συνεργασία που εξελίσσεται και συνεχίζεται και πιστεύω απολύτως ότι θα εξακολουθήσουμε να είμαστε στρατηγικοί εταίροι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλα και πρόεδρο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χασβήλη. Συνάδελφοι, έτσι ολοκληρώνουμε τη συζήτηση αυτή. Το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τους συγκεκριμένου μας προσκεκλισμένους για την πολύ ενδιαφέρουσα ενημέρωση που λάβαμε για τη συνεργασία με τρίτες χώρες σε αποστολές και πα παρουσίαση τρόπων βελτίωσης της συνεργασίας αυτής. Κυρία Κάνσλαντα, υπολογίζουμε σε τακτική ενημέρωση από πλευρά σας. Να είσαστε βέβαιοι λοιπόν ότι θα το ξαναβάλουμε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη, παρουσιάζοντας ενδεχομένω και άλλους εταίρους. Να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ και θα ήθελα να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί τους πανελίστες μας. Και παρακαλώ να παραμείνετε στην αίθουσα για να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Yes, I hope can uh, actually.